μα κάθε φορά τι εξελίξει, ενδεχομένω και οι ισπανικέ αερογραμμέ κάποια στιγμή να αρχίσουν μια απεργία. Επομένω, δεν γίνεται για του λόγου αυτού να αναβάλουμε κάθε φορά την ψηφορία. Πρέπει να προχωρήσουμε τη μερίσια διάταξη. Δεν υπάρχουν έγγραφα αυτή τη στιγμή, αλλά όχι μόνο στη δική μας συνεδρίαση και στι υπόλοιπε συνεδριάσεις των Επιτροπών δεν υπάρχουν έγγραφα. Θα σας διαβάσω λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Προβλέπεται ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Έχουμε επίσης ένα σχέδιο έκθεσης το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και έχουμε επίσης μια έκθεση από την κυρία Μπαντία Κουτσέτ όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση του 2010, εφαρμογή του προγράμματος εργασίας και στη συνέχεια έχουμε και την έκθεση του κ. Μόρτεν Λόκιγκάρτ για τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων που θα κάνουμε σήμερα. Είναι μια απλή εισαγωγή για τι εκθέσει που θα δούμε αργότερα. Και έχουμε επίση και μια συνεδρία συντονιστών σήμερα και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε πλήρη, πλήρη φακέλου με τα έγγραφα. Δυστυχώ, όπω σα είπα, καμία επιτροπή δεν κατάφερε να λάβει έγγραφα για τις ε, σημερινές συνεδριάσεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά, μάλλον όχι, δεν τα έχουμε καν μπροστά μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Δεν τα έχουμε διαθέσιμα. Φαντάζομαι θα τα δείτε αύριο το πρωί και θα καταφέρουμε να συζητήσουμε αύριο εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο. So,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 θα έχουμε μία ακρόαση όσον αφορά τα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Carl Schmitt, στην αίθουσα 1α2, στο άλλο κτίριο. Πρόκειται για μια ακρόαση λοιπόν και αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μια πιο μεγάλη αίθουσα, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες. Πορτογαλικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα. Έχουμε Μαλτέζικα στη Δερμηνία, αλλά για ποιο λόγο δεν έχουμε Βουλγαρικά. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, σας διαβάζω, λέει πρόεδρος, τις γλώσσες που δεν έχουμε διαθέσιμες στη Δερμηνία. Έχουμε λοιπόν όλε τι γλώσσε από τα βουλγαρικά, τα πορτογαλικά, τα σλοβανικά, τα εσθονικά, τα λιθουανικά, τα Λετουνικά και τα μαλτέζικα. Μου φάνηκε λίγο περίεργο ότι είχαμε, να είχαμε Μαλτέζικα μάλλον, γιατί δεν έχουμε βουλευτή από τη Μάλτα. Αύριο θα έχουμε όλες τις γλώσσες εργασίας εκτός από τα Σουδικά, τα αστωνικά, τα Λουθανικά, τα Λετωνικά και τα Μαλτέζικα. Αυτά όσον αφορά τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Ας περάσουμε στην πρώτη ψηφοφορία. Δύσκολη θα έλεγα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν με τον ακόλουθο τρόπο. προκειμένου να καταφέρουμε να καλύψουμε και τις επόμενες δύσκολες ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τρούπελ, πρωτού ξεκινήσει η ψηφοφορία. Έλγα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Όσοι συμμετείχαν στην δουλειά για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Βασικά, κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, καθώ επίση και τα μέλη τη Γραμματεία, καθώ επίση και όλου του υπόλοιπου οι οποίοι συνέβαλαν στην έκθεση αυτή. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια η οποία έγινε. Γίνανε κάποιε πολύ καλέ συζητήσει. Συζητήσαμε πάρα πολύ το θέμα της ψηφιακής βιβλιοθήκης για την Ευρώπη και θελήσαμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να καταστήσουμε το σχέδιο αυτό, ένα σχέδιο το οποίο θα γνωρίσει επιτυχία και το σχέδιο αυτό της ε, ψηφιακής βιβλιοθήκης για την Ευρώπη πραγματικά μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία για την Ευρώπη και μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, σταθμό και ορόσημο για την πολιτιστική πολιτική της Ευρώπης. Από πολιτικής πλευράς υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Είδαμε ότι ε, ανακύπτουν, αν θέλετε, κάποιες ε, πρώτες ε, ευίωνες στάσεις, αλλά θα θέλαμε να σημειωθούν περισσότερες βελτιώσεις στο μέλλον, όχι μόνο σε επίπεδο κοινοτικό, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί η κατάλληλη ευρωπαϊκή βούληση και επίσης να καταφέρουμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τους πολίτες για το σημαντικό αυτό σχέδιο, το κοινοτικό σχέδιο της ε, Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Νομίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στο σημαντικότατο αυτό σχέδιο για την πολιτιστική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, νομίζω ότι και από χρηματική πλευρά πρέπει να δούμε αν τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να συμβάλλουν και αν θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε και από τον κοινοτικό προπολογισμό. δηλαδή το σχέδιο αυτό θα καταφέρει να έχει τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς πόρους. Κάτι τέτοιο είναι απολύτω απαραίτητο, ιδίως στα πλαίσια τη νέα στρατηγική τη ε, Λισαβόνα. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, σαφώς χρειαζόμαστε χρήματα, χρειαζόμαστε πόρους και οι πόροι αυτοί θα πρέπει να διατεθούν στα πλαίσια της νέας στρατηγικής. Επίσης, στα πλαίσια της έκθεσης μιλάμε για την ευρωπαϊκή κληρονομιά, η οποία δεν προστατεύεται πλέον από το copyright. Επομένως, είναι δυνατό για πάρα πολλά πνευματικά έργα πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφιοποιηθούν προκειμένου να γίνουν ε, διαθέσιμα για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για όλους τους ανθρώπους αστικά που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το σχέδιο της ψηφιακής βιβλιοθήκης θα είναι ένα σχέδιο στο οποίο θα καταφέρουν να συμμετέχουν ε, όλοι οι πολίτες που το επιθυμούν. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διευθετήσουμε και το ζήτημα των πνευματικών αυτών έργων που ακόμα καλύπτονται από copyright. Ενδεχομένω να πρέπει τα έργα αυτά να γίνουν διαθέσιμα με κάποιε συγκεκριμένε προποθέσει υπό ένα συγκεκριμένο σύστημα όρων που θα πρέπει να καλύπτονται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή, ποιο σύστημα πληρωμή θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να έχει κανεί πρόσβαση στα έργα αυτά. Νομίζω ότι και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να διαπαιτηθούν προκειμένου το εγχείρημα αυτό τη ψηφιακή βιβλιοθήκη να στεφθεί με επιτυχία. Σαφώ δεν θα θέλαμε εδώ πέρα να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη σαν αυτή του Google, όπου στην αρχή διαφημίστηκε ως μια εντελώ ανοιχτή ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπου όλα τα έργα ήταν προσπελάσιμα και προσβάσιμα και λίγο αργότερα συνειδητοποίησαμε ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Το ζήτημα αυτό θα μα απασχολήσει και του επόμενου μήνε. Έχουν υποβληθεί πολλέ τροπολογίε. Επί της αρχής όμως πρέπει να πω ότι στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας κάναμε μια πολύ χρήσιμη, πολύ καλή συζήτηση και από τη στιγμή που θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε και τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην έκθεση αυτή, θα καταφέρουμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα έχει πραγματικό πολιτικό βάρος και θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε περισσότερο το σχέδιο αυτό προς τα έξω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι συμμετέχοντες στην έκθεση αυτή και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τις πληροφορίες. Ε, κύριε Σμίτ, δεν έχουμε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Απλώς πρέπει να περάσουμε... Σας παρακαλώ, ακούστε με. Η κυρία Τρούπερ παρουσίασε συμβιβαστικέ τροπολογίε με το σκιώδη συγητή. Και εν συνεχεία γίνανε αυτές οι προφορικέ τροπολογίε και δεν θα δεχτώ, δεν θα τις δεχτώ παρά μόνο εάν η εισηγήτρια τις δεχτεί, τις προφορικές τροπολογίες, εντάξει, καταλάβατε. Διότι αυτό αφορά διάφορες πολιτικές ομάδες. Λοιπόν, προφορικές τροπολογίες δεν θα γίνουν δεκτές εκτός εάν η κυρία Τρούπελ τις έχει αποδεχθεί. Έχουμε μία προθεσμία για τις τροπολογίες. Όποιος παραβεί την ε, προθεσμία αυτή, εντάξει, να το σκεφτώ. Αλλά σήμερα αυτές οι προφορικές ε, τροπολογίες που δεν θα γίνουν απαδεκτές θα μπορούσαν να ακουστούν στην Ολομέλεια από την πολιτική του ομάδα και να υποβληθούν εκεί. Λοιπόν, έχουμε στην Επιτροπή συμφωνήσει μία προθεσμία υποβολής και πρέπει να την ε, σεβαστούμε για να μην διαταράξουμε και την συμβιβαστική εργασία της εισηγήτριας. Άρα λοιπόν μπορούν αυτές να υποβληθούν από την ομάδα στην ε, Ολομέλεια. Θα υπάρξει από πλευράς ε, ΕΛΚ μία ξεχωριστή ψηφοφορία, ένα split vote σε μια συμβιβαστική τροπολογία. Το ζητήσατε αλλά δεν γίνεται. Μόνο αν γίνει αποδεκτή η ψηφοφορία, η τροπολογία, συγγνώμη, μπορείτε να, να ζητήσετε εν συνεχεία ξεχωριστή ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Εάν περάσει σήμερα, μπορείτε εν συνεχεία να ζητήσετε ξεχωριστή ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Σήμερα όμως όχι. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Παράγραφος 1, τροπολογία 24 της κυρία Φερχάιεν, Wir müssen zählen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer ist dagegen? Κατά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abgelehnt. Απορρίπτεται. 25. Έχει αποσυρθεί. Παράγραφος 1α, τροπολογία 26, ξεχωριστή ψηφοφορία ζητήθηκε για την πρώτη παράγραφο. Υπέρ, κατά, δεκτή. Δεύτερη παράγραφος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1β, 27, υπέρ, κατά, Αποχές δεκτή. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29 Κύριο Γκάλο υπέρ. Κατά. Ευχαριστώ. Δεκτή. 30. Τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. Η προφορική τροπολογία της κυρίας Βεζιάτ δεν έγινε δεκτό προς ψηφοφορία γιατί η κυρία Τρούπολ δεν το επισημεί. Προχωρούμε στην 31. Βεζιά υπέρ. Κατά. Πρέπει να μετρήσουμε. Υπέρ παρακαλώ. Σηκώστε το χέρι σας. 12. Yeah, you can. Zwölf. So. 12. Κατά. 3, 4, 5, 6. Angenommen. Δεκτή. Είμαστε στην 32. Υπέρ. Κατά. Κανείς αυτή η επόμενη τροπολογία δεν έχει γίνει αποδεκτή, καθότι προφορική. Προχωρούμε στην 33, Βριζιά, Ταβάρες, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 34, υπέρ, κατά, δεκτή. 35, υπέρ, κατά, δεκτή. 36, υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 39. 39. Υπέρ. Κατά. Για, για να ελέγξουμε. Ε, να μετρήσουμε και πάλι. Υπέρ. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also alle von uns. Wer ist dagegen? 13. 7, 8, 9, 10. Angenommen. Δεκτή. 13 υπέρ 10 κατά. Δεκτή. 38. Dagegen? Κατά. Δεκτή. 40 υπέρ κατά, δεκτή. Συμβιβαστική α, ε, <laughs> υπέρ, κατά, από, ε, εγκρίνεται, δεκτή. 41 καταπίπτει προφορική τροπολογία από την εισηγήτρια. Ε, προφορική τροπολογία 3. Υπέρ, Α, ε, έχει καλυφθεί η προφορική 3. Ε, προχωράμε στο 43. Υπέρ, κατά, χες, δεκτή. 44. Υπέρ. Κατά. χες, δεκτή. 46. Υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. Προφορική τροπολογία 4. Η Εισηγείται υπέρ. Ε, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 45 έχει αποσυρθεί. 47 παράγραφος 9. Σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα, πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 48, υπέρ, κατά, δεκτή. Η προφορική τροπολογία δεν τη δεχόμαστε γιατί η κυρία Τρούπελ την απορρίπτει. 49, τροπολογία 49, υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά απορρίπτεται 51 υπέρ κατά πρέπει να μετρήσουμε υπέρ είναι 12 του ΕΛΚ και ένας απέναντι 13 κατά 10, 11, 12. 13 κατά. 13-13 απορρίπτεται. 52. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτη, πρώτο τμήμα, παρακαλώ, δεκτό. Ε, υπέρ κατά δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά Απο, απο, ε, απορρίπτεται. Το πρώτο τμήμα δεκτό, το δεύτερο απορρίπτεται. 54. Υπέρ, κατά, δεκτή. 54, ε, δύο τμήματα. Το πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα του 54, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεκτό και το δεύτερο τμήμα. 55. Πρώτο τμήμα. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος απορρίφθηκε. 55 δεύτερο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται 56 έχει αποσυρθεί η ψη... Κύριε Κάβαντα, προχωράμε στο 57. Προφορική τροπολογία δεν έγινε δεκτή. 57 υπέρ. Κατά. Πρέπει να μετρήσω. Υπέρ παρακαλώ. Μετράμε. Alle 13 von, wie viel haben wir? 12 oder 13 dürfen wir haben? 12. Also die 12 EVP. Und weiter? 13, 14. Dafür. Υπέρ ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, δεκτή. 59 υπέρ, κατά, δεκτή. 60 υπέρ, κατά, δεκτή. 61 υπέρ, κατά,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 Wer ist dagegen? Κατά. Απορρίπτεται. 62 έχει αποσυρθεί. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 65 έχει αποσυρθεί. 66 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 68 δεκτή, 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, Wie bitte beim nicht. Können wir noch mal sagen, wer ist dafür? Ξαναψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ και μετράμε. 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Dagegen waren 14, 12. 14 zu 12. 14 έναντι 12. Αποσύρεται. Ε, συγγνώμη, ε, απερίφθη. Η επόμενη έχει αποσυρθεί, 72. Απορρίπτεται 73 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ε, συμβιβαστικές Β. Συμβιβασμός Β δεν μπορούμε να ψηφίσουμε με ξεχωριστή ψηφοφορία, ψηφίζουμε κανονικά υπέρ ή κατά. Υπέρ, παρακαλώ, συμβιβασμός Β. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71. Τι κάνουμε τώρα με την παράγραφο 18, εκτός μικροφώνου όμως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 Δεκτή. 79 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 82 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 83 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 86 υπέρ όχι, το, η 84 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε 86 υπέρ κατά δεκτή. 85 υπέρ κατά δεκτή. 87 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά δεκτό. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 90 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά Άποχες. Απορρίπτεται. 99 έχει αποσύρθει. 92 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή. 93 έχει αποσύρθει. 94 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Γίνεται δεκτή από την εισηγήτρια η προφορική τροπολογία της κυρίας Σάκε. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. 95. Κυρία Σάκε. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Πάμε στην 96. Υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ένα. Υπέρ. Κατά. Δεκτό. Δύο είναι ε, τα εκτιμώντας. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τρία υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Πέντε σε δύο μέρη. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο, υπέρ, κατά, Άποχες, δεκτό, έξι, υπέρ, κατά, ε, ξανά παρακαλώ, υπέρ, υπέρ, κατά, άποχες, δεκτό, εφτά, έχει αποσυρθεί, οχτώ, υπέρ, εννέα, ε, συγγνώμη, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 9. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία αυτή, η προφορική δεν γίνεται δεκτή. Τροπολογία 11. Ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ κατά ε, πρέπει να μετρήσουμε τη 10, το 10 υπέρ Υπέρ παρακαλώ, υπέρ ψηφίζουμε τώρα. Υπάρχει πρόβλημα? 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16. Ωραία, δεκτεί. 12, Σάκε, υπέρ. Είναι dagegen. Κατά. Können wir noch einmal. Wer ist dafür? Επαναλαμβάνουμε. Υπέρ. Δεκτή. Δεκτή. Δεκατρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβασμός Χ. Περίεργο αυτό το Χ. Λέει η πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη 18. Κάβαντα. 18. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική 9 δεν γίνεται δεκτή. Προχωράμε στη 17. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 19 υπέρ, κατά, δεκτή. Ξανά παρακαλώ. 19 υπέρ, κατά ε, απορρίπτεται 23 υπέρ υπέρ 23 παρακαλώ κατά απορρίπτεται στο Ιανόφ 20 υπέρ κατά δεκτή 21 υπέρ κατά Δεκτή. Τώρα έχουμε την ε, γνωμοδότηση της ε, Γιούρη. Ε, ένα υπέρ κατά δεκτή. Δύο υπέρ κατά δεκτή. Τρία υπέρ κατά πρέπει να μετρήσουμε. Υπέρ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sind 14. So, 14. Wer ist, der, wer ist äh... Κατά, παρακαλώ. Νομίζω ότι ξεχάσατε να μετρήσετε δύο ψήφους στο Προεδρείο. Είχα, είχατε τρεις ψήφου από το Προεδρείο. Μία υπέρ, δύο κατά. Για να ξαναψηφίσουμε και ο κύριος Γραμματέας θα μετρήσει. Υπέρ την τροπολογία 3 της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Την 3 παρακαλώ, υπέρ. 16 λοιπόν. Δεκτεί λέει η πρόεδρος, Δεκτεί. 4 υπέρ, κατά, Δεκτεί. 5 υπέρ, κατά, Δεκτεί. 6 υπέρ, δεκτεί. 7 υπέρ, κατά, δεκτεί. 8 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 9 υπέρ, δεκτή. 10 υπέρ, κατά, δεκτή. Η γνωμοδότηση τώρα η, της Ήτρε. Τι να κάνω με το, την ασυμβατότητα με την παράγραφο 1. Α, αφήνουμε την 1, ψηφίζουμε την 2. 2 παρακαλώ, υπέρ. Κατά δεκτή. Ε, η 3 καλύπτεται από το εκτιμώντας G παράγραφος 5. Προχωράμε στο, 4 υπέρ. Κατά αποχές ε, δεκτή. 5 υπέρ κατά δεκτή. 6 υπέρ κατά δεκτή. 7 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, η 10 καλύπτεται από το, τις παραγράφους που αναφέρει εκεί στα εκτιμούντας. 10, όχι μάλλον τις παραγράφους 5, 17 κτλ. Απορρίπτεται η 10, 11 υπέρ, κατά, δεκτή. Η 11 δεκτή. 12 υπέρ κατά απορρίπτεται. 13 καλύπτεται από άλλες ε, παραγράφους, ε, από άλλες, 13 υπέρ, δεκτή, ε, 13 καλύφθηκε, το 14 δεκτή, 15 δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά δεκτή, 18 υπέρ κατά δεκτή, 19 υπέρ κατά δεκτή, 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α υπέρ κατά αποχές δεκτή, β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ωραία. Τελική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές ομόφωνα δεκτή η έκθεση και συγχαίρουμε σερμά την εισηγήτρια κυρία Τρίπελ wir kommen jetzt zum Bericht des Kollegen. Και τώρα προχωρούμε στην έκθεση του κυρίου Σόριν Ιβάν. Καθορισμός νέας ψηφιακής ατζέντας για την Ευρώπη από το 2010 στο digital.eu. Να αρχίσουμε. Έχετε τα έγγραφά σας, κύριε Κύριε Σόριν, Ιβαν, έχετε κάτι να προσθέσετε, αν θέλετε, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που κατέθεσαν και γιατί βοήθησαν ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είμαι πεπισμένος ότι η τελική της μορφή θα είναι κάτι στο οποίο θα συζητήσουμε όλοι ε, το υλικό το οποίο προέκυψε από τη συζήτηση αναλύθηκε και ε, αναπτύχθηκε. Δεν έχω και πολλά παραπάνω να πω. Ε, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και ελπίζω να πάνε όλα καλά στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και αρχίζουμε με την παράγραφο 1, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Δεκτή. Δύο. Υπέρ. Α, πρέπει να πάμε στη 10. Πολύ ωραία. Προχωρούμε στη 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και οι 70 είναι ταυτόσιμοι, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 11 και 71 triple, behind, είναι επίσης ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές. Δεκτές. Προχωράμε στην 4, στην 5, συγγνώμη, 5 του κυρίου Μάτουλα. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6 υπέρ, κατά, θα ήθελα να παρακαλέσω το ΕΛΚ να συμμετάσχει στην ψηφοφορία όπως θέλει, υπέρ, κατά. Ή, επαναλαμβάνουμε, το 5, τροπολογία 5, Γιώργη Μάτουλα, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6, υπέρ, κατά, Αποχές δεκτή. 7. Έχουμε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Πρώτο, δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, άποχες, δεκτό. 8. Υπέρ. Κατά άποχες δεκτή. Προχωρούμε στο 12. Τρίπελ υπέρ, 12, ε, 12, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 56, 13 ε, και 73, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι, συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Η ε, ξεχωριστή ψηφοφορία από την ΚΟΕ ζητήθηκε 13, 73. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό, Δεύτερο, υπέρ κατά αποχές δεκτό. 14 και 16 είναι ταυτόσιμες υπέρ, 14 και 60 συγγνώμη, κατά αποχές δεκτές, 15 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 18 ε, και 46 ψηφίζουμε υπέρ, κατά αποχές δεκτές. 19 υπέρ, κατά δεκτή. Χαίρομαι, ήταν και δική μου. 23 υπέρ. Υπέρ, 23, ψηφίζουμε. Α, όχι. Δεν χρειάζονται όλα οι επόμενες. Και προχωρούμε στην 26. 26 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ κατά απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 33 είπε κατά αποχές δεκτή. θα, δεχτείτε την τροπολογία της κυρίας Κώστα, ρωτάει πρόεδρος τον εισηγητή. Τότε τη διαβάζω. Είναι προφορική που θα γίνει δεκτή από τον εισηγητή. Και λέει, τροπολογία 34. τονίζει την σημασία της ε, πρόσβασης ε, των ε, λιγότερο προνομιούχων ή των μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων στην ψηφιακή τεχνολογία και στις καινοτομίες, της τεχνολογίες αυτές που χρειάζονται για μια κοινωνική ανέλυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας και εισηγείται ειδικά προγράμματα όπως παρένθεσης ή inclusion ε, τεχνολογία, κλείνει παρένθεση, τα οποία προγράμματα θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις ομάδες. Μα τι γίνεται, μπορείτε να μου το πείτε αυτό. Η τροπολογία δεν είναι όλα αυτά που διάβασα. Α, τζάμπα έκανε τον κόπο, λέει η κυρία Πακ. Λοιπόν, είναι μία μικρή προσθήκη που λέει στην παρένθεση, λέει, ή inclusion, και η τροπολογία προσθέτει and existing technology. And existing technology κλείνει η παρένθεση. Αυτές τις τρεις λεξούλες λοιπόν προσθέτει η τροπολογία. Κανένας δεν είναι κατά. Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική αυτή τροπολογία. Assistive and assistive technology, λέει η παρένθεση. Λοιπόν, υπέρ κατά, αποχές δεκτή. 35. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 45 υπέρ κα... κατά αποχές Δεκτή. Ήταν και δική μου, λέει η πρόεδρος. 47. 47. Και 48, 49, 50 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, ε, δεκτές. 52 υπέρ. Α, προχωρούμε στην 55. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 61 τώρα υπέρ υπέρ κατά πρέπει να μετρήσουμε. Υπέρ, παρακαλώ. Αν τη Yeah, it's okay. It's enough. the Liberals for It's Δεκτή. Εξήντα έξι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Εξήντα εφτά. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, δεκτή. 69 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και ψηφίζουμε ολόκληρη την τροποποιημένη έκθεση υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτεί, Συγχαίρω τον εισηγητή. Και προχωρούμε στην επόμενη έκθεση του Ιβου Μπέλετ. Ε, το θέμα είναι διακυβέρνηση του ίντερνετ, τα επόμενα βήματα. Μήπως κύριε Μπέλετ θέλετε να προσθέσετε κάτι, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ε, ε, να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας προς το στόχο μας να αυξήσουμε την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διακυβέρνηση του παγκόσμιου διαδικτύου. Να ευχαριστώ ίσο πολύ για τη συνεργασία, για τις τροπολογίες. Αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπής είναι η Επιτροπή Ήτρε. Είμαι και εγώ μέλος ε, στην Επιτροπή και θα κάνω προφανώς ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προασπίσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού στην Επιτροπή Ήτρε. Yeah. Είναι πάντα καλό αν όταν φοράμε δύο καπέλα σε δύο επιτροπές. Παράγραφος 1, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 έχει αποσυρθεί. 4 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. εκτός μικροφώνου. Α, το, η προφορική ψηφοφορία βρίσκεται στην, στο πίσω μέρος της σελίδας, σελίδα 2 της Marie Christine Verziat. Στην παράγραφο 1, παράγραφος 1, ε, και εκεί λέει προφο, προφορική τροπολογία, ο συγητής είναι υπέρ, ναι, είναι υπέρ, οπότε εντάξει. 7, ε, τροπολογία 7. Πρώτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8, τροπολογία 8, υπέρ, κατά, αποχές, αποχές δεκτή. 9, ο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13 σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, υπέρ, κατά, υπέρ, κατά, αποχές, δεύτερο μέρος υπέρ, Κατά. Αποχές. Δεκτό. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκτή. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί 19, 21. Όχι. Όχι. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχ... αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 νίξ 24 υπέρ Μα δεν λέει τίποτα στην 23 λέει η πρόεδρος Α, καλά, 23 υπέρ κατά υπέρ παρακαλώ ξανά την 23 υπέρ κατά Δεκτή. 24 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Ψηφίζουμε ο, ολόκληρη τροποποιημένη έκθεση υπέρ κατά κατά παρακαλώ κατά αποχές ομόφωνα δεκτή Συγχαίρουμε τον Ιβο Μπέλετ. So, jetzt kommen wir zum äh, τώρα έχουμε το γενικό της Trüppel. Μία σύντομη παρατήρηση λέει έχω λάβει υπόψη μου όλες τις τροπολογίες, διότι τις θεώρησα ότι βελτιώνω σημαντικά το κείμενο πλην από δύο του κυρίου Μπίσκι, τις οποίες ε, δεν δέχτηκα, όχι για ιδεολογικούς λόγους και για λόγους αρχής, αλλά για λόγω του περιεχομένου ε, ζητούν οι δύο τροπολογίες, διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία δεν έχουν θέση εδώ στην έκθεση αυτή. Άρα λοιπόν απέρριψα τις δύο τροπολογίες αυτές μόνο για το περιεχόμενο, όχι για άλλους ιδεολογικούς λόγους. Πολύ ωραία η πρόεδρος. Ψηφίζουμε. Το, ε, ένα, τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές. Ξανά παρακαλώ την 2 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πέντε υπέρ κατά αποχές δεκτή. Very briefly, I would like to propose to the colleague. Πολύ σύντομα θα ήθελα να προτείνω ε, στους συναδέλφους από το ΕΛΚ να απόσχουν τις 6 και τις 7, να μην ε, καταψηφίσουν. Μήνυμα ελίτ. Ε, 6 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, δεκτή, δεκτή, δεκτή. Μπίσκι, η τοπολογία, λέει η πρόεδρος. Ωραία. Θέλω να πω, η κυρία Τρούιπελ έχει δίκιο. Εδώ πρόκειται για απαλλαγή, όχι για να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Δεν πρόκειται για το τι ζητάμε για τον επόμενο προϋπολογισμό, αλλά αφού το ζητήσατε όλοι, εντάξει, δεν λέω ότι έγινε μεγάλη ζημιά που κάνουμε αυτό το λάθος, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα ψηφίζουμε ολόκληρη την τροποποιημένη έκθεση της κυρίας Τρουιπέλ υπέρ, κατά, κατά παρακαλώ, αποχές, Ο, δύο αποχές. Με δύο αποχές έγινε δεκτή, σας συγχαίρω κυρία Τρουιπέλ. So, damit haben wir Ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν αυτά τα τεχνικά θεματάκια, τα οποία βέβαια είναι ουσιώδη. Και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση της κυρίας ε, Μαρία Μπάντια Μπάντια-Ικούτσετ. Κάθε δύο χρόνια από το Συμβούλιο και την Κομισιόν συντάσσουμε μια κοινή έκθεση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα προγράμματα κατάρτισης. Και αυτά τα προγράμματα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικά διότι εστιάζουν στις δεξιότητες κλειδιά τις οποίες έχουμε ήδη αποφασίσει. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα εντονότατα διότι ολόκληρη η στρατηγική της Λισαβόνας δεν ε, θα αξίζει τίποτα εάν δεν προσέξουμε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σας ε, προτείνω λοιπόν να μελετήσετε ενδελεχώς την έκθεση αυτή. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση και παρακαλώ την εισηγήτρια να μας ε, παρουσιάσει την πολύ σημαντική αυτή έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω τις ε, σημειώσεις μου στα αγγλικά, γι' αυτό λοιπόν θα τα πω στα αγγλικά σήμερα. Όπως είπε και η Πρόεδρος, έχουμε μία έκθεση για την πρόεδρο των ε, ε, εκπαιδευτικών ε, πολιτικών και της κατάρτισης κατά το 2008-2009. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη της και, ε, στρατηγικές και τεχνικές διαβίου μάθησης και προσπαθούμε να κάνουμε την επαγγελματική και πανεπιστημιακή κατάρτιση πιο δελαστική και να αυξήσουμε την ανώτερη εκπαίδευση. Μιλάμε για ευκαιρίες οι οποίες ε, θα μας δώσουν νέες διοξιότητες για νέες πρωτοβουλίες. Η ανακοίνωση προτείνει και μία σειρά από μέτρα για να προχωρήσουμε, την, ε, να δώσουμε μια όθηση στον τομέα αυτό. Και δίνει και μία εικόνα της ε, τρέχουσας κατάστασης. Η έκθεση σχεδίου της ε, εκθέσεως προόδου ε, καθορίζει ποιοι είναι οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι κατά τα τελευταία χρόνια και για τις βασικές αρμοδιότητες λέει ότι έχει γίνει αρκετή σημαντική πρόοδος ε, στο σχολικό πρόγραμμα και κάποιες χώρες έχουν δημιουργήσει πολύ συγκεκριμένε στρατηγικέ και προγράμματα δράσης για να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες, κυρίως για τη γραφή και ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Και επίσης ε, προάγεται επιχειρηματικότητα μέσω συγκεκριμένων στόχων, όπως για παράδειγμα εταιρικέ σχέσεις μέσω επιχειρήσεων και ε, ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ε, διοικούμε μικροεπιχειρήσεις. Τώρα, για τη διαβίου μάθηση, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένες στρατηγικές διαβίου μάθηση και έχουν γίνει προσπάθειε για να υποστηρίξουμε την ευέλικτη ε, ε, εκπαίδευση. Για την επαγγελματική κατάρτιση, η προσαρμοστικότητα των συστημάτων έχει αντιμετωπιστεί ως τμήμα της διαδικασίας της Κοπεχάγης και οι περισσότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δώσει προτεραιότητα στο ο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας. Τώρα, για την ανώτερη εκπαίδευση έχουμε όλο και μεγαλύτερη γνώση στις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η μεγαλύτερη γνώση και η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση είναι θεμελιώδου σημασία για τις ε, στρατηγικές διαβίου μάθησης. Έτσι έχουν υιοθετηθεί μέτρα για να μπορέσουν να ενταχθούν και τα ε, μικρότερα, κατώτερα στρώματα κοινωνικο-οικονομικά. Η έκθεση λέει ότι παρόλα αυτά απαιτούνται και άλλες βελτιώσεις. Η ανακοίνωση επισημαίνει την ανάγκη να ενισχύσουμε την καλύτερη στάση μας προς την περαιτέρω ε, εκπαίδευση και είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα η ψηφιακή δεξιότητα, η δυνατότητα του να μαθαίνει κάποιος μέσω της μάθησης και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την επιχειρηματικότητα και την πολιτισμική γνώση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ε, δεξιοτήτων για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης και για την ε, εκπαίδευση των ενηλίκων. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ε, βασικών δεξιοτήτων. Πρέπει να δοθούν επίσης μεγαλύτερες προσπάσεις για τη γνώση γραφής και ανάγνωσης και τις μειονεκτούσες ομάδες και θα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης απόδοσης ε, για τις δυνατότητες ανάγνωσης και επίσης ε, μια καλύτερη προσέγγιση μάθησης για τις ε, ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προγράμματα συγχρονισμός της ανώτερης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Επίσης, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των ε, δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας και αναμένεται να αυξηθούν τα προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Στενή συνεργασία επίσης πρέπει να υπάρχει και με τον κόσμο των επιχειρήσεων και είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο για να έχουμε πιο ελκυστικές προσόντα και κυρίως δυνατότητες κινητικότητας για τους φοιτητές. Για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει επένδυση από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας τρόπος για να έχουμε περαιτέρω χρηματοδότηση. Θα πρέπει να επεκταθεί η εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημοσίου τομέα και θεωρούμε ότι οι εταιρικέ ε, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλους τομείς, κυρίως του τομέα ε, του χώρου της εργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει αυτή η έκθεση να χωριστεί σε διάφορα εκπαιδευτικά στάδια. Πριν από δύο χρόνια είχαμε μία έκθεση η οποία έγινε από την κυρία Νόβακ και ήταν έτσι διαρθρωμένες οι ιδέες και αυτό ε, θα μας δώσει ένα πιο σαφές κείμενο γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες γιατί μου φάνηκε ότι ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο αυτό που θέλαμε να πούμε. Θα ακολουθήσω λοιπόν τη δική της την άγουσα. Θα ήθελα τώρα να θέσω ένα ερώτημα το οποίο ίσως θα πρέπει να θέσουμε όλοι στους εαυτούς μας. Οι δε, βασικές δεξιότητες είναι οι σωστές, είναι οι δεξιότητες που πρέπει να αξιολογήσουμε. Η εκπαίδευση των διδασκόντων είναι πολύ σημαντική για μένα. Θα πρέπει να αυξηθεί η κινητικότητα, θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν να μετακινηθούν και να έχουν τη δυνατότητα να πάνε από τον ένα χώρο στον άλλον. Από δημοσιεύματα στον τύπο και από εκθέσεις θα δείτε ότι οι δάσκαλοι δεν χρησιμοποιούν όλα τα προγράμματα τα οποία εγκρίνουμε εμείς για την κινητικότητά τους. Ε, ίσως δεν υπάρχει χρόνος ή ίσως αυτά τα προγράμματα δεν τα έχουμε σκεφτεί καταλήλως για τη δική τους κινητικότητα. Θα πρέπει να τα βελτιώσουμε λοιπόν όλα αυτά. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νέες θέσεις εργασίας. Μιλάμε για νέες δεξιότητες, για νέες θέσεις εργασίας, αλλά δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι νέες θέσεις εργασίας. Εάν δεν ξέρουμε λοιπόν ποιες είναι, δεν ξέρουμε και πώς θα ε, επιμορφώσουμε τους ε, καθηγητές, αλλά και πώς θα μορφώσουμε τους φοιτητές. Ως προς τα κριτήρια τώρα, νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την εμπειρία μας, αλλά και την οτροπία που έχουμε όλοι ως προς τη γνώση. Για τις μειονεκτούσες ομάδες, η παιδεία θα πρέπει να θεωρείται ως ένα μέσο ενσωμάτωσης, ως ένα μέσο καταπολέμησης της ένδυας και φυσικά θα πρέπει ε, να καταπολεμήσουμε και το φαινόμενο όλων αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο πολύ νωρίς. Ε, σε πολλές χώρες είναι πρόβλημα αυτό και στην χώρα μου επίσης. Ε, το θέμα των επενδύσεων εξετάζεται μόνο για το μέλλον. Πολλές φορές η παιδεία ε, διαφεύγει της ε, πολιτικής των κρατών μελών. Δεν είναι κάτι στο οποίο απλώς διαθέτουμε κονδύλια και έχουμε αποτελέσματα αμέσως. Είναι κάτι το οποίο είναι μακροπρόθεσμο και πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν ε, το γνωρίζουν αρκετά αυτό. Νομίζω ότι το κόστος της μηδενικής δράσης στον τομέα αυτό θα είναι καταστρεπτικό για όλους μας. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση των ελληνικών και τη διασύνδεσή της με τη διαβίου μάθηση, θα πρέπει τα χρόνια της εμπειρίας θα πρέπει να ενταχθούν στο παραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης. Όλοι χρειάζονται δυνατότητες για να μεθαίνουν και ε, οι ενήλικες που δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, σύμφωνα με μία έρευνα της Eurostat, είναι κατά 23% λόγω οικογενειακών ευθυνών και είναι κατά 22% ως αντικρουόμενο με το πρόγραμμα εργασίας. Το κόστος είναι το τρίτο πιο σημαντικό εμπόδιο που δεν επιτρέπει στους ενήλικες να συμμετέχουν σε, θέματα, σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίση, χρειαζόμαστε νέε δεξιότητε για νέε θέσει εργασία, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και αυξημένη κινητικότητα. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα πιο πολύ όλα όσα μαθαίνουμε στην αγορά εργασία. Και αυτό είναι θεμελιώδου σημασία για, την, ε, ε, για τους νέους επαγγελματίες και τις δυνατότητές τους για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Ε, θέσεις εργασίας για το μέλλον. Επαναλαμβάνω, ποιες θέσεις εργασίας για το μέλλον. Πράσινες, λευκές, μπλε θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους, διότι πολλές από τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα, από, τις εργασ... από τα επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα, θα εξαφανιστούν. Ε, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να διασυνδεθούν πολύ πιο στενά με την αγορά εργασίας, χωρίς να ξεχνάμε ε, και συγκεκριμένες μελέτες, ε, διαφοροποίηση του, των επαγγελματικών μας δεξιοτήτων δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, ψηφιακές γνώσεις, νέοι τρόποι εργασίας. Επίσης, αρκεί η τρέχουσα συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθούν. Από ό,τι φαίνεται, στο τελευταίο Συμβούλιο Παιδείας, κάποια κράτη-μέλη έθεσαν την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας. Κάτι το οποίο είναι καλή ιδέα φυσικά. Βρισκόμαστε στο 2010, μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της, ένδυσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού και αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε και την παιδεία προς αυτό το στόχο. Του χρόνου, το 2011, θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού σημαίνει ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες είναι ένας τρόπος άτυπης παιδείας και θα έχουμε ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και περαιτέρω δεξιοτήτων και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ως δεξιότητες για νέες ε, θέσεις εργασίας και ε, να θεωρούνται και ως ε, επίσημη εκπαίδευση. Αυτά λοιπόν είναι όλα όσα σκέφτηκα, διάβασα και νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα πρέπει να τα περιλαμβάνει. Βέβαια, με τα χαράς θα μπορούσα να ακούσω τους περισσότερους από εσά και να έχουμε νέες ιδέες, προτάσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αγαστά μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ε, Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε πολύ καιρό για συζήτηση το πολύ 45 λεπτά. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακουστούν οι ιδέες μας, γιατί η Μαρία τον Μάρτιο, 22-23 Μαρτίου, θα παρουσιάσει την έκθεσή της και καλό θα ήταν να συμπεριλάβει ορισμένε ε, ιδέες από τα μέλη μας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς ε, δεξιών μου. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Πρέπει να σας πω ότι η ανακοίνωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική, μία από τις σημαντικότερες στον τομέα της εκπαίδευσης και το συμπέρασμα, το πόρισμα της έκθεσης αυτής θα μπορούσε να αποτελεί τελικά ένα είδος οπισθοδρόμησης όσον αφορά την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν κατάφεραν να πετύχουν τους βασικούς μας στόχους και τα τελικά αριθμητικά στοιχεία είναι αρνητικά. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ πέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι από κοινού θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή έκθεση για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θα μιλήσω ουγγρικά και θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, το ζήτημα του media literacy, το να μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς τα νέα μέσα επικοινωνίας. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βομβαρδιζόμαστε από πάρα πολλέ νέε πληροφορίε, από πολλού νέου διάβλους επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να προωθήσουμε το ζήτημα αυτό του γραμματισμού, του media literacy, της ικανότητας των πολιτών να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν τις δεξιότητες αυτές οι πολίτες και επίσης θα πρέπει σωματικά και ενδεχομένω να χαμογελάσετε, αλλά θα πρέπει και σωματικά οι πολίτε μα να βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση. Δηλαδή, να... η φυσική του κατάσταση να είναι καλή. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανισορροπία στην ζωή του. Να εργάζονται, για παράδειγμα, 10 ώρε και να μην εξασκούνται σωματικά καθόλου. Νου υγιή εν πνεύμα υγιή ουσιαστικά. Το έχω πει αυτό και στο παρελθόν, ενδεχομένω να σα κάνω να χαμογελάτε, αλλά νομίζω θα πρέπει να περάσει και η ιδέα αυτή στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Du denkst sicher an den Sport und da stimmen wir dir alle zu. Σίγουρα, σίγουρα έχει στο νου σου το σπορ και όλοι συμφωνούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα είπα προσωπικώς και στην κυρία Μπαντίε Κούτσετ, αλλά το θέμα της παιδείας ε, εμένα με απασχολεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι να διευκολύνουμε την κινητικότητα των ε, καθηγητών και δασκάλων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτή την κινητικότητα, να είναι μεγαλύτερο το δέλεαρ του να μπορεί να διδάσκουν διάφοροι καθηγητές σε διάφορες χώρες. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μου φαίνεται σημαντικό. Και επίσης τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την εκμάθηση των διαφόρων ξένων γλωσσών, ευρωπαϊκών γλωσσών στα σχολεία, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν από μικρά. Ε, αυτά τα σημεία θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Ευχαριστώ. Καταρχά να ευχαριστήσω τη συναδελφό μα για τι πολύ καλέ ιδέε που μα παρουσίασε και να αφαιρθώ σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Αναφερθήκαμε σε όλα αυτά τα ζητήματα εκπαίδευση και κατάρτιση και σε όλα αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο. Υπάρχει όμω ένα σημαντικό πρόβλημα δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δεξιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλες αυτές τις απαιτήσει. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν κανείς θέλει να στεφτεί το όλο εγχείρημα με επιτυχία, θα πρέπει να υπάρχει κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη. Και μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο και βρισκόμαστε και στα μέσα μια οικονομική κρίση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο προπολογισμό των κρατών μελών δεν είναι ο ευκταίο. Επομένω υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα χρηματοδότησης, πώς θα καταφέρουμε ουσιαστικά να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση και την έρευνα. Μέρος λοιπόν της εκθεσής σας θα πρέπει να φέρετε στο πώς θα καταφέρουμε να συσχετίσουμε καλύτερα το κοινοτικό και το εθνικό επίπεδο. Πώς θα καταφέρουμε να έχουμε κάποια κοινά συμφέροντα, κάποιους κοινού στόχους, πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε κοινέ πολιτικές και πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε κοινού στόχους. Και πέρα από την δημοσιονομική πτυχή των πραγμάτων θα πρέπει να δούμε επίση και πώ μπορούμε να προσεγγίσουμε από πολιτική πλευρά με κοινό τρόπο το ζήτημα της εκπαίδευση και πώ θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τρόπο του ίδιου του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτέ. Πώ θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια σημαντικά ζητήματα, τα βασικότερα ζητήματα, πώ θα καταφέρουμε να εναρμονίσουμε τα εκπαιδευτικά μα συστήματα, πώ θα καταφέρουν αυτά να ευθυγραμμιστούν με τι νέε απαιτήσει που έχουν ανακύψει και πώ θα καταφέρουμε ουσιαστικά να εξομοιώσουμε τα εκπαιδευτικά μα συστήματα, να έρθουν όλα στο ίδιο υψηλό επίπεδο. Η κυρία Κώστα, παρακαλώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισαγωγική της παρέμβαση, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρης. Θα ήθελα να επισημάνω τρία πράγματα. Πρώτον, τα θέματα τα οποία θέτουμε εμείς, όπως κάνει και η ανακοίνωση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, η εκπαίδευση και οι στρατηγικές εναντίον της οικονομικής κρίσης και οι στρατηγικές της ε, Ευρώπης ε, για το 2020 θα πρέπει να βαθυνθούν περισσότερο για να ξέρουμε γιατί δεν καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2010. Αυτό το οποίο φαίνεται να προχώρησε μόνο είναι το θέμα των ε, πτυχίων σε επιστημονικούς τομείς, σε φυσικές επιστήμες. Αλλά υπάρχουν ακόμα μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού και μεγάλη έλλειψη ε, δεξιοτήτων ακόμα και στις φυσικές επιστήμες. Θα πρέπει να έχουμε και κάποια καινοτόμα στοιχεία για στόχους τους οποίους δεν έχουμε συμπεριλάβει. Συμπερίζομαι πάρα πολύ το θέμα των διδασκόντων. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα θα ήταν ίσως ε, μη Επιτροπή να εμβαθύνουμε και στο θέμα αυτό και να κάνουμε μία σύγκριση ως προς τον τρόπο κατάρτισης και επιμόρφωσης στη, στη διάρκεια του διδακτικού τους βίου και να δούμε και τι έκαναν οι χώρες οι οποίες έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα στο θέμα αυτό. Επίσης, το θέμα της... Ε, μουσικής και πολιτιστικής παιδείας δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα μπορούσε να βοηθήσει και τα διάφορα συστήματα εκμάθησης ε, για τα νέα παιδιά και επίσης θα πρέπει να δούμε πόσο έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός ε, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για θέματα πανεπιστημιακά και έρευνας. Σε πολλές χώρες και στη δική μου τα τελευταία χρόνια περικόπηκε ο προϋπολογισμός και ίσως εδώ θα πρέπει να δεσμευτεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά και εμείς για να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό. Και ένα τελευταίο σημείο είναι το πού βρισκόμαστε ως προς τη δυνατότητα σύγκρισης του συστήματος ε, ECOF, το Equal Quality Framework, δηλαδή συγκρισιμότητα και ε, κατά πόσον υπάρχει και κυκλοφορία των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Κάποιες χώρες είναι ακόμα πίσω στα θέματα αυτά, ίσως θα πρέπει να γνωρίζουμε λίγο καλύτερα πώς έχουν τα πράγματα και να ε, γίνει και μια ενημέρωση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και ανώτατη εκπαίδευση, όχι μόνο εντός των πανεπιστημίων, αλλά και ανταλλαγή μεταξύ πανεπιστημιακών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Και εδώ συμμερίζομαι και τις ιδέες της ε, Μαρία Μπαντιέ Κουτσέτ. Κλείνοντας να πω ότι το Συμβούλιο Υπουργών μου φαίνεται ότι πράγματι μίλησε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παρά το σεβασμό της αυτονομίας των εκπαιδευτικών συστημάτων, θα πρέπει να πάμε πέρα από το σύστημα του ανοιχτού συντονισμού και να αρχίσουμε να έχουμε ένα πιο κοινό όραμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για κατευθυντήρες γραμμές, αλλά θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο περαιτέρω, διότι πλέον ως προς τους στόχους, ως προς τα σχολικά προγράμματα και στα αποτελέσματα της κατάρτισης, και της εκπαίδευση θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα σύγκριση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λίγο πιο συνεκτικοί σε σχέση με αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο συζητάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα των πολιτών μας στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το πανεπιστήμιο. Το αναφέρατε αυτό, αλλά θα ήθελα να πω και το εξή. Όταν τα πανεπιστήμια μας δεν καταφέρουν πλέον να ακολουθήσουν το αμερικανικό παράδειγμα και να εμπλακούν περισσότερο ουσιαστικά με το τομέα τη έρευνα, τότε οι επενδύσει μα πηγαίνουν χαμένε. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει και τα πανεπιστήμια μα να εστιάζονται περισσότερο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Επίση, κάποια βασικά προγράμματα κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε από πώ μπορούμε και συγκεκριμένε τομεί του πληθυσμού να του κατευθύνουμε προ συγκεκριμένε δεξιότητε. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από διάφορε έρευνε ότι οι γυναίκε είναι πάρα πολύ δυνατέ σε συγκεκριμένου τομεί. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο τέτοια προγράμματα. Επίση, πολλέ φορέ ε, εκπαιδεύουμε και καταρτίζουμε πολίτε χωρί να λαμβάνουμε υπόψη μα τις απαιτήσεις της ε, αγοράς εργασίας. Με αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί να καταλήγουν άνεργοι στο τέλο. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου λοιπόν ποια είναι η προσφορά στην αγορά εργασία και πώ θα πρέπει εμεί να προσαρμοστούμε στι απαιτήσει αγορά εργασία. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό, η επιτυχία αυτή έχει υποτιμηθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει επίση να υπάρχουν μέσα κοινά για όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, όπου υπάρχουν ακόμα κάποιοι διαθέσιμοι πόροι. Νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό και θα καταφέρει να καταστήσει, πιστεύω, το, την έκθεσή μα το πρόγραμμά μα πολύ πιο αποτελεσματικό. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται μια ε, σαφής αναφορά στα αθλήματα στην έκθεση αυτή. Στην έκθεση μέχρι στιγμής δεν αναφερόμαστε καθόλου στις αθλητικές δεξιότητες. Γιατί είναι και αυτές δεξιότητες που θα μπορούσαν να είχαν πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να φερθεί κανείς στον τομέα αυτό και να τον περιγράψει σωστά, αλλά αν όντω περιλαμβάνει το αθλητισμό στον στρατηγική τη Λισαβόνα, τότε νομίζω ότι και στην έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνουν οι δεξιότητε που συνδέονται με τον αθλητισμό. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μπαντία Ικουτζέτ ε, για την πολύ σημαντική αυτή πρώτη προσέγγιση του ζητήματος. Ε, είναι περισσότερο μια αγωνία αυτό που εκφράζω παρά ε, κάτι παραπάνω αναρωτιέμαι αν σε αυτή την έκθεση και αν στην πρόταση που θα κάνουμε εμείς ε, θα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω μία ενότητα πεδίων εκπαιδευτικών που δεν αναφέρονται πουθενά ίσως γιατί δεν σχετίζονται άμεσα με την αγορά εργασίας. Θα το δούμε και αύριο αυτό το πράγμα με την σχέση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Το ζήτημα σε αυτή την έκθεση είναι να τονίσουμε μόνο τις δυνατότητες ε, σχέσεις έρευνας ή επιστήμης με αγορά εργασίας ή μήπως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας γενικότερες απαιτήσει μιας κοινωνίας που ε, δεν θα έλεγα ότι καλύπτεται μόνον από την ε, ανάγκη για μια επαγγελματική αποκατάσταση. Από την άποψη αυτή, πέρα από τον αθλητισμό, θεωρώ ότι σε αυτή την έκθεση θα πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί η σημασία των ανθρωπιστικών σπουδών δεν είναι δυνατόν να αποσυνδέουμε την εκπαίδευση με την έννοια της παιδείας όμως, education or culture, από τις ε, ανθρωπιστικές σπουδές. Ακόμη και αν δεν πρόκειται να είναι το εργαλείο μέσα από το οποίο θα βρουν μια... Ε, ε θα, θα αναπτύξουν περισσότερα προσόντα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εκτιμώ ότι χωρίς τις ανθρωπιστικές σπουδές δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η Ευρώπη. Και ένα άλλο στοιχείο που επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι στην προσπάθεια για να ε, ομογενοποιήσουμε, ίσως να φέρουμε πιο κοντά τα διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης, νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθεθεί η ανάγκη στα προγράμματα τα εκπαιδευτικά να προσθεθούν και μαθήματα ιστορίας της Ευρώπης. Εκτιμώ ότι μόνο ε, με μια τέτοια προσέγγιση όπου θα ο κάθε λαός, κάθε εθνικό κράτος θα έχει την υποχρέωση να διδάσκει την ιστορία των άλλων 26 κρατών ή όσων θα προκύψουν στην πορεία, μόνον έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε και την προσέγγιση την πολιτιστική, την πολιτισμική ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη και να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Συνοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση και με την διδαχή της ιστορίας και βεβαίως να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη των ανθρωπιστικών σπουδών στην επαγγελματική κατάρτιση. Χωρίς αυτές φοβάμαι ότι θα έχουμε μια τεχνοκρατική προσέγγιση που δεν νομίζω ότι είναι το μοντέλο που θα θέλαμε να έχουμε για μια Ευρώπη του άμεσου μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μερικές παρατηρήσεις να θυμηθούμε όλοι εδώ ότι ακροβατούμε. Οι δεξιότητες κλειδιά, τις οποίες η Κομισιόν εφεύρευε και τις οποίες δεχτήκαμε, είναι ουσιαστικά προτάσεις που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Είναι προτάσεις. Και η Κομισιόν πήρε αυτή την πρωτοβουλία την οποία θέλαμε και συνεχεία ε, συνέχισαν και άλλοι φορείς αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα στην διδακτέα ύλη, ούτε μπορούμε να προδιαγράψουμε τι θα μάθει ποιος. Ούτε η Κομισιόν μπορεί να το κάνει. Αυτές οι δεξιότητες κλειδιά τις ονομάσαμε, τις ε, παρουσιάσαμε, πείσαμε το Συμβούλιο να τις δεχτεί το Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει να σεβαστεί αυτή την ε, δέσμευση και να τις ε, μετατρέψει σε πολιτική. Η έκθεση τώρα πρόκειται κυρίως, εστιάζει την προσοχή της κυρίως στην υλοποίηση αυτών των στρατηγικών για την εξέλιξη των δεξιοτήτων κλειδί. Αυτό που πρέπει να κρίνουμε είναι τι έκαναν οι χώρες, ε, τα κράτη-μέλη για να ε, εφαρμόσουν αυτές τις, ε, την ανάπτυξη και να διευκολύνουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Δεν μπορούμε τώρα να παρουσιάσουμε προτάσεις ή να ζητήσουμε από τη Μαρία να συμπεριλάβει τα πάντα, ό,τι είναι στην καρδιά μας, δηλαδή σε αυτήν την έκθεση. Αν και εγώ συμμερίζουμε τη γνώμη των περισσότερων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού. Όμως αυτό δεν είναι δεξιότητα κλειδί. Βεβαίως, όπως και η κυρία Καντάν το έχει ήδη προδιαγράψει, θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού, των καθηγητών, των δασκάλων. Επίσης, το θέμα της ε, των μέσων ενημέρωσης και της αξιοποίησης των γνώσεων. Αυτό επίσης μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως ε, για παιδιά 8 με 11 ετών. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω. Και το άλλο θέμα που θα συζητήσουμε αύριο, το θέμα της ε, συνεργασίας ε, μεταξύ λυκείων και πανεπιστημίων. Και αυτό έχει άμεση σχέση με τον εξυγχρονισμό των ε, λυκείων, της γυμνασίων και λυκείων. Για να δούμε πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε την ε, διδακτέα ύλη με θέματα τα οποία συνάδουν ε, με την οικονομική και βιομηχανική πολιτική. Και ένα άλλο θέμα, το ανέφερε ο κύριος Μπόρις, έχουμε ήδη κάνει μια προσπάθεια ε, εξομοίωσης ε, των ε, πανεπιστημίων. Η διαδικασία της Μπολόνιας δεν είναι τίποτα το διαφορετικό. Σε αυτό αποσκοπεί. Είπατε να μην μιμηθούμε ένα αμερικανικό μοντέλο. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν έχω πολύ υψηλή γνώμη για το αμερικανικό μοντέλο. Εγώ θέλω να προωθήσουμε το δικό μας ευρωπαϊκό μοντέλο και πιστεύω ότι ακολουθούμε ήδη μια σωστή πορεία. Αυτά ήθελα να πω επί του θέματος και εν κατακλείδη. Η Κομισιόν και εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πατήσει παρθένο έδαφος με αυτές τις δεξιότητες κλειδί. Και έχουμε προχωρήσει, έχουμε πραγματικά ξεκινήσει αυτές τις καινοτομίες και γι' αυτό πιστεύω ότι η έκθεση της Μαρίας είναι εξαιρετική. Η κυρία Χάνιμπολ έχει ζητήσει το λόγο. Thank you, Chair. Um, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ μαζί σας. Οι συζητήσεις αυτές, οι εκθέσεις αυτές είναι σίγουρα αρκετά δύσκολες. Δεν είναι εύκολο να οριοθετήσει κανείς τα πράγματα πολύ εύκολα. Εμείς κάνουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση, αν θέλει, του ζητήματος, χωρίς όμως να καταφέρνουμε πάντα να το οριοθετήσουμε πλήρως. Υπάρχουν κάποια σαφή σημεία στην έκθεση αυτή. Είναι καλό το ότι αναφερόμαστε στι βασικέ δεξιότητε. Και νομίζω ότι η έκθεση αυτή αναφέρεται πολύ καλά σε αυτέ τι δεξιότητε και τι αναλύει. Όμω, δεν αναφέρεται στην ε, πρόοδο. Δίδονται κάποιοι γενικοί όροι που δεν μας βοηθούν όμως και πάρα πολύ. Και πραγματικά πρέπει να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε με την έκθεση αυτή στα πλαίσια της Επιτροπής. Θέλουμε τα πράγματα να μείνουν στάσιμα ή θέλουμε ουσιαστικά περισσότερες πληροφορίες. Γιατί δεν ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με την ε, διαδικασία της Μπολόνια η διαδικασία της Μπολόνια είχε να κάνει ουσιαστικά με αυτόνομα πανεπιστήμια τα οποία θα συνεργάζονταν μεταξύ τους. Ενώ από ό,τι φαίνεται τώρα ασχολούμεθα μεμονωμένα με τα εκπαιδευτικά συστήματα κάθε κράτους μέλους και ουσιαστικά λέμε ότι ορισμένα πράγματα θα θέλαμε να γίνουν από τα κράτη-μέλη, ότι θέλουμε να αναλάβουν κάποια δράση. Δεν έχουμε όμως εδώ πέρα ένα απολογισμό για κάθε, κράτες, κάθε κράτος μέλος. Έχουμε μια γενική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα το οποίο καθιστά την όλη συζήτηση ασαφή, αόριστη. Εγώ νομίζω ότι τα όσα λέγονται για τις βασικές δεξιότητες είναι πολύ θετικά και δεν διαφωνώ με τις προτάσεις που ακούστηκαν να προσθεθούν δηλαδή και άλλες δεξιότητες. Απλώς αμφιβάλλω για το τι δρόμο ακολουθούμε αυτή τη στιγμή, για το πού θα, καταλή... θα καταλήξουμε και τι θέλουμε να πετύχουμε. Αρχικά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε καλύτερα τα πράγματα και να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε αυτή την έκθεση. Καλό θα ήταν αν γνωρίζαμε ποιο κράτος μέλος έκανε ποιο πρόγραμμα, τι έκανε, πότε και πώς. Ε, θα είχαμε μία επισκόπηση έτσι της κατάστασης. Αλλά τα στοιχεία αυτά δεν θα μας τα δώσει το Συμβούλιο, ούτε η Κομισιόν θα μας τα έδινε, ακόμα και να τα είχε. Ωραία θα ήταν αυτή όμως, να είχαμε μια γενική επισκόπηση. Ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Παλιατέλη. Παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ε, And there ε, ε, Στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μου, υπάρχει ένα τμήμα του Πανεπιστημίου που μόλις τελείωσε μία έκθεση για την επαγγελματική κατάρτιση. Εχθέ δημοσιεύτηκε, αν δεν την έχετε μπορούμε να σας αποστείλουμε. η δημοσίευση. Αν την έχετε, μια χαρά και νομίζω ότι εκεί έχετε πάρα πολλά πληροφορίες για το πρόβλημα το οποίο ανέφερε η κυρία Χάνιμπολ. Ναι, αλλά πρόκειται μόνο για την επαγγελματική κατάρταση, έτσι δεν είναι. Δεν είναι για τα benchmarkings, για τα συγκριτικά προγράμματα, είναι τα, της επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά και οι άλλοι τομείς είναι πολύ σημαντικοί. Σας ευχαριστούμε όμως για την υπόδειξη αυτή. Παρακολουθούμε βεβαίως ε, και τις εξελίξεις και τις εκθέσεις του ΣΕΝΤΕΦΟ ε, από πολύ κοντά. Ε, θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στην, εκτελεστική, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως μπορείτε να μας πείτε τι έχουν κάνει ορισμένες χώρες και τι δεν έχουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω από την τελευταία σας παρατήρηση. Αυτό το οποίο έχετε εδώ στα χέρια σας στηρίζεται στις εθνικές εκθέσεις, οι οποίες είναι λεπτομερώς διατυπωμένες. Παράλληλα λοιπόν ε, με τις εκθέσεις ε, αυτές ε, και δεδομένου ότι η ανακοίνωσή μας είναι πάρα πολύ σύντομη, έχουμε κάνει εμείς διάφορες συγκριτικές μελέτες για κάθε χώρα βάσει αυτών των εθνικών εξέσεων. Με πολύ προσοχή προχωρήσαμε και με πολύ προσοχή διατυπώσαμε και με συνένεση βεβαίως με τα κράτη-μέλη. Έχουμε τους, τα στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία ένα κράτος μέλος, ορισμένα σχόλια ε, του τι έγινε στο συγκεκριμένο κράτος μέλος και όσοι θέλετε να το κοιτάξετε αναφέρομαι στο έγγραφο εργασίας ε, στον τίτλο ε, της ανακοίνωσης. Εδώ πρόκειται για βασικές δεξιότητες για τη διαβίωμαση, όχι για τη σχολική εκπαίδευση μόνο. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να προετοιμάσουμε τα, τους μαθητές των σχολείων για το τι θα επέλθει εν συνεχεία πέραν των σχολείων. Και επίσης ε, καλύπτει και τους, ε, την εκπαίδευση ενηλίκων όπως είπε και η κυρία Μπαντία, στην ε, σχολική, στο σχολικό πλαίσιο έχουν σημειωθεί πολύ ικανοποιητικές εξελίξεις. Βεβαίως πολλά έχουμε ακόμα να κάνουμε. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης ε, του διδακτικού προσωπικού. Επίσης πρέπει να βελτιώσουμε περισσότερο την πρόσβαση των μειονεκτούντων ομάδων και δεδομένου ότι αυτές οι βασικές δεξιότητες είναι αρκετές, ε, πρέπει για κάθε μία να διαπιστώσουμε τι εμπόδια πρόσβασης και κατάρτισης υπάρχουν, πού υπάρχουν ελλείψεις. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις τις οποίες έχει δεχθεί ε, και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δώσει το έναυσμα ε, ε, πολλών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Έτσι ξεκίνησαν λοιπόν, έδωσαν μια όθηση Δεδομένου ότι δεν αναφερόμαστε εδώ σε εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρογνώμονες σε ορισμένους τομείς, εδώ αναφερόμαστε στο μέσο όρο βασικών ικανοτήτων, είναι πολύ σημαντικό να ξεκινούν παράλληλα πολλές πρωτοβουλίες. Και τέλος, ενώ μιλούμε ε, για την εκπαίδευση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η εκπαίδευση ε, συνδέεται άμεσα με την οικονομία, τον οικονομικό τομέα, την οικονομική ανάπτυξη ε, έχουμε και ε, το, πρόγραμμα 2020 ε, με το οποίο συνδέεται όλη η στρατηγική δηλαδή αυτή και οι παράλληλοι τομείς συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τόιτσε, λέει πρόεδρος. Μπορώ να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Ο κύριος Σμιτ. Σας ευχαριστώ, συγγνώμη που δευτερολογώ. Άκουσα ότι τα πράγματα είναι πολύ ε, δύσκολα, ότι βρισκόμαστε στην κόψη του, ξη, του ξηραφιού. Ότι έχουμε εντοπίσει κάποιε δεξιότητε, αλλά δεν ξέρουμε τελικά τι συνέχεια να δώσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω, γιατί στην Ουγγαρία, αν κάποιο θέλει να βρει μια δουλειά, θα μπορούσε να απευθυνθεί σε πάρα πολλέ επιχειρήσει όπω η Deutsche Bank, η Siemens, η Nokia. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάρη στην ε, παγκοσμιοποίηση μπορεί κανείς να εργαστεί στις εταιρείες αυτές. Από την άλλη, απορούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν κάποιες βασικές δεξιότητες. Από τη στιγμή που μιλάμε για την ελεύθερη κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία τόσο ατόμων όσο και κεφαλαίων, πιστεύω ότι και οι νέοι, οι πολίτες, θα πρέπει να είναι απαραίτητα σωστά προετοιμασμένοι. Μαρία. Κυρία Μπαντία Κουτσέτ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι αδύνατον με όλη αυτή την πληθώρα πληροφοριών και προτάσεων να απαντήσω σε όλους έναν προς έναν. Ε, πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, διότι εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η έκθεση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και με ικανοποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι διαπιστώνω ότι και εσείς συμμερίζεστε το ενδιαφέρον μου. Νομίζω ότι συμμερίζομαι και όλες τις ιδέες που ακούστηκαν εδώ. Εδώ στην Επιτροπή μας συνήθως είμαστε πεπισμένοι ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες. Συνήθως δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα. Αν όμως στεκόμασταν σε αυτό δεν θα μπορούσαμε να εργαστούμε πάνω σε τίποτα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες μας. Όταν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και μπορούμε να προσφέρουμε νέες ιδέες και συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, νομίζω ότι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρονται γι' αυτό και με τον τρόπο τους όταν μπορούν και όπως μπορούν το εφαρμόζουν. Θεωρώ λοιπόν ότι η δυνατότητα που μας δίνεται αυτή τη στιγμή είναι να εργαστούμε πολύ καλά, να ετοιμάσουμε μια πολύ καλή έκθεση και εάν είμαστε και λίγο δημιουργικοί, ε, αυτή τη στιγμή που χρειαζόμαστε τη δημιουργικότητα, ε, να έχουμε και μία έκθεση η οποία θα είναι δημιουργική και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα το κάνει το Συμβούλιο όλο αυτό που θα ετοιμάσουμε. Να σας ευχαριστήσω όμως όλους για τις προτάσεις σας και ελπίζω από τις προτάσεις σας ε, θα έχω και τις ανάλογες τροπολογίες στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ θέμα του Μόρτεν Λόκεγκάρτ είναι «Δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωση, δημιουργία μια δημόσια σφαίρα στην Ευρώπη». Πιστεύω ότι αν σκεφτείτε σε τέσσερα χρόνια θα έχουμε πάλι ευρωπαϊκές εκλογές, θα πρέπει να ομολογήσετε ότι δεν έχει πανευρωπαϊκή συζήτηση για πανευρωπαϊκά θέματα. Κανένας δεν είναι καλύτερος Ευρωπαίος από τον άλλον. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε ε, και, τους, και τη δημοσιογραφία και τα μέσα ενημέρωσης να κάνουν τις ανταποκρίσεις τους λίγο πιο ευρωπαϊκές και από πλευράς δηλαδή εθνικών πολιτικών. Είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα λοιπόν μία έκθεση με τέτοια θέματα, μέσα ενημέρωση και δημοσιογραφία. Ο κύριο Λέκεγκάρτ έχει το λόγο. Θα συνεχίσω στα αγγλικά. Πρέπει όμω να είμαι συγκεκριμένο, επομένω θα μιλήσω δανέζικα. Φορέστε παρακαλώ τα ακουστικά σας. Minister uddannelse. Øh, mine Κύρια Πακ, πολύ σωστά είπατε ότι εγώ είμαι δημοσιογράφος και ε, η πολιτική μου πείρα είναι πολύ σύντομη. Όμως, έχω γράψει για την πολιτική στις εφημερίδες της χώρας μου, της Δανίας. Έχω κάνει Έχω κάνει εκθέσεις από το Κοινοβούλιο. Ε, το, η δουλειά μου δηλαδή ήταν να κάνω πολιτική ανταπόκριση από το Κοινοβούλιο της Δανίας. Πολύ συχνά ασχολήθηκα και με την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχόλιά μου ήταν είτε θετικά είτε αρνητικά ανάλογα με την περίσταση. Στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος στον οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε τα ευρωπαϊκά ζητήματα, τα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή της κοινή γνώμης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ανέλαβα να εκπονήσω την παρούσα έκθεση και ε, στόχος μου είναι να συζητήσω και με πολλούς ενδιαφορομένους του κλάδου. Εδώ και 50 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό οικοδόμημα το οποίο έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία, έχει καλύψει πάρα πολλές πτυχές της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών Και ναι, μεν πολλές φορές ε, τα δημοψηφίσματα ή οι ευρωεκλογές ε, δεν ε, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Ευρωπαίοι πολίτες φαίνεται να ρίχνουν το ηθικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση, για περισσότερη επικοινωνία. Και αυτή είναι και η πρώτη μου παρατήρηση. Όσον αφορά τώρα τα προγράμματα. Κατά την άποψή μου, οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι και ενημερωμένοι ως προς τα θέματα που συζητάμε και όλα αυτά που ψηφίζουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη ε, και αυτό προκύπτει και από την πείρα μου ως δημοσιογράφος. Όπως αυτό που θα σας πω και μόλις τώρα. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να κάνει το οτιδήποτε, να επικοινωνήσει, να δημοσιοποιήσει κάτι με κάθε κόστος οι πολίτες ε, είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ενδιαφερθούν ε, σε κάποιο βαθμό και για τα όσα αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί να δούμε πόσο ε, ανοιχτός, πόσο εύκολο είναι να κάνει κάποιος προπαγάνδα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία 60 χρόνια διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθεί μια νέα νοοτροπία. Και εδώ έρχομαι και στην επόμενη πτυχή. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου γίνονται πάρα πολλά πράγματα εδώ στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν πολλές καλές προθέσεις, πολλά καλά προγράμματα, αλλά στα κράτη-μέλη ανακύπτουν προβλήματα. Στα κράτη-μέλη δεν υπάρχει κατάλληλη γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να παρακινήσουμε τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν, να μορφώνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο στον οποίο οι ευρωπαϊκές υποθέσεις θα είναι θέμα καθημερινής συζήτησης σε κάθε χώρα μέλος όπως ε, είναι θέμα καθημερινής συζήτησης τα όσα συμβαίνουν εντός της χώρας, η μικροπολιτική της ε, πόρο απέχει από τη σημερινή πραγματικότητα. Οι πολίτες θα πρέπει να θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά θέματα, οι ευρωπαϊκές υποθέσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής τους. Δεν μπορούμε να πείσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρονται μόνο στα ευρωπαϊκά θέματα. Εγώ έχω εντοπίσει κάποιους τομείς, τους οποίους θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις πρώτος ο παραδοσιακός πολιτικός τομέας, ο αγνός πολιτικός τομέας, όπου είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες ε, κατά κάποιο τρόπο στο ευρωπαϊκό σύστημα, στο σύστημα ε, λήψης δημοκρατικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πολιτικό χώρο και χώρο συζήτησης ε, για την κοινή γνώμη. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, στο Ευρωπαϊκά Συμβούλια δεν ναι, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προς αυτή την κατεύθυνση. Στους πολίτες δεν υπάρχει ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται στο Συμβούλιο και αυτό είναι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα. κατ' εμέ σε κάποιες περιπτώσεις δεν φτάνουν, όπως και εδώ, δεν φτάνουν όλα τα στοιχεία τα οποία ε, λαμβάνουμε από κάθε πρωτεύουσα, αλλά αντίστοιχα υπάρχει το αντίστροφο πρόβλημα. Όσα συζητάμε εμείς εδώ δεν φτάνουν κατά ανάγκη σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Στις ευρωπαϊκές υποθέσεις λοιπόν θα πρέπει να συμμετέχουν και τα κράτη-μέλη από την αρχή μιας διαδικασίας λήψης απόφασης. Δεν θα πρέπει να ε, λειτουργούμε ο καθένας ξεχωριστά και να τους αποκόπτουμε από τις διαδικασίες. Εγώ σκέφτομαι τη χώρα μου για παράδειγμα, τη Δανία ως ε, παράδειγμα όλων αυτών που σας είπα και έχω σκεφτεί ε, τι ακριβώς θα μπορούσαμε να κάνουμε για να έχουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ ημών και βουλευτών ε, στο Κοινοβούλιο της Δανίας, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξελών και Κοπενχάγης. Αυτό θα το αναφέρω και στην έκθεσή μου. Και μπορώ να σας πω ότι αυτή τη φορά, σε αυτή τη θητεία για παράδειγμα, δεν μας ε, χαροποιεί καθόλου το γεγονός ότι ο, επίτροπος, ε, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, δεν όρισε και έναν αρμόδιο επίτροπο για θέματα επικοινωνίας. Αυτό θα απέστελνε ένα πιο στεναρό μήνυμα για την επικοινωνία και τη δημοσιοποίηση των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Βέβαια αυτό θα συνεχίσει να συζητάτε και κάτι ακόμα το οποίο για μένα είναι σημαντικό είναι το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτά καθ' αυτά. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Δεν έχω καμία πρόθεση και καμία ψευδέστηση ότι μπορούμε και θα πρέπει να παρισφρήσουμε στην ελευθερία των ε, ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε μέχρι τούδε και να σας πω εδώ ότι και εμείς ως φιλελεύθεροι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν μια σειρά ευρωπαϊκών θεμάτων τα οποία δεν συζητιούνται. Αυτό είναι και πολιτικό πρόβλημα, αλλά είναι και πρόβλημα μέσω μαζικής ενημέρωσης. Και είναι και παράδοξο, διότι όπως σας είπα, ναι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουν όπως θέλουμε εμείς, αλλά Εξετάζοντας λίγο την κατάσταση στα κράτη-μέλη, διαπίστωσα ότι στη Γερμανία, για παράδειγμα, ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, το BBC, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, δεν ε, ε, λαμβάνει τα διάφορα ευρωπαϊκά θέματα όσο σοβαρά θα έπρεπε. Στη Δανία έχουμε δύο κρατικά ε, κανάλια και θα θέλαμε σε αυτά τουλάχιστον να συζητιούνται περισσότερο τα ευρωπαϊκά θέματα. θα μπορούσαμε να αποστείλουμε και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Το ξέρω ότι η θητεία του Άμστερνταμ προστατεύει, η εντολή συγγνώμη, του Άμστερνταμ προστατεύει την εθνική επικουρικότητα σε τέτοια θέματα. Αλλά εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες συστάσεις για μηνύματα που θα μπορούσαμε να αποστείλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τώρα τον, την έντυπη δημοσιογραφία, νομίζω ότι οι εφημερίδες ε, κάνουν καλύτερη πληροφόρηση, αξιοπρεπή αν θέλετε. Ε, νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στη βελτίωση της ενημέρωσης από, ε, τους, ε, από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους νέους τρόπους επικοινωνίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ εμείς στην Επιτροπή μας επαναλαμβάνουμε πάρα πολύ συχνά. Πρόκειται για πληροφόρηση η οποία πολύ συχνά ταξιδεύει μέσω διαδικτύου ή ε, τα λεγόμενα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα νέο κόσμο και είναι λίγο δύσκολο ακόμα και να προβλέψουμε πώς θα αναπτυχθεί όλο αυτό το δίκτυο. Εγώ το συζήτησα και με, την, ε, ε, και με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής Για πρώτη φορά το Κοινοβούλιο βρίσκεται και στο Facebook, επομένως ε, είχαμε και διάφορες ενδιαφέρουσες εμπειρίες, βρισκόμαστε σε μια πειραματική φάση Οι επισκέψεις ε, της ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου είναι περίπου 1.500. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πολύ ικανοποιητικό. Προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αλλά αυτά τα νέα μέσα επικοινωνίας όπως το Twitter και το Facebook θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. γνωρίζουμε ότι και στις Βρυξέλλες λαμβάνονται πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Εμείς που εργαζόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι πολίτες. Υπάρχει και η δορυφορική τηλεόραση, υπάρχει ένα, μια ολόκληρη στρατιά, αν θέλετε, δημοσιογράφων παρόντων εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά δεν αρκούν για την κατάλληλη ε, ενημέρωση. Χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση, κατάλληλη παιδεία και ε, χρειάζεται να δείξουμε ότι το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλο αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι ε, εδώ σε αυτή την πρώτη μου παρέμβαση μπόρεσα να σας παρουσιάσω τα ουσιαστικά σημεία και νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα μπορούσε να πει και την άποψή της ε, και για προβλήματα τα οποία θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό. Και Υπάρχει κάτι το οποίο θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Δεν θα καθαριστερήσω άλλο σήμερα τη συζήτηση, αλλά φαντάζομαι ότι στην επόμενη συνεδρία που θα συζητήσουμε το θέμα θα μπορέσω να σας παρουσιάσω αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να προσπαθήσουμε να επικοινωνούμε με τους πολίτες και με νέα μέσα. Αυτά λίγο πολύ λοιπόν για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πρέπει όμως να υπάρχει ένα πρόγραμμα επικοινωνίας από πλευράς θεσμικών οργάνων. Και ναι μεν εγώ θεωρώ ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά ολοκληρωμένο, ένα σύστημα ολοκληρωμένο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το γεγονός ότι θα θέλαμε και έναν αρμόδιο ad hoc επίτροπο επί του θέματο, αρμόδιο επί του θέματος και δεν ξέρω αν τα πράγματα θα προχωρήσουν το ίδιο καλά χωρίς ένα αρμόδιο επίτροπο. Στην προηγούμενη θητεία, όπω ξέρετε, υπήρχε η κυρία Βάλστρομ, η οποία ήταν αρμόδια για θέματα επικοινωνία. Αυτό για μένα ήταν προεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και χάρη στο έργο της ε, προήθηκε η συνεχή συνεργασία ε, κυρίως με, τους, ε, με τα περιφερειακά τελεοπτικά δίκτυα υπήρχε μια συνεχής ροή πληροφοριών αλλά συμμερίζομαι λίγο και τις επικρίσεις που έγιναν στην Επίτροπο Βάλστρομ ότι έκανε λίγο παραπάνω προπαγάνδα πώς έπρεπε. Στο μήνυμα το οποίο περνούσε, δεν υπήρχε ποτέ καμία επίκριση, καμία κριτική και φαινόταν σαν ε, προπαγάνδα. Αυτά λοιπόν είναι τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να αποστείλουμε. Σαφώς υπάρχει πάρα πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό και δεν θα ήθελα εγώ να κάνω προπαγάνδα, σας το είπα αλλά καλό θα ήταν να ενημερώνουμε περισσότερο. Οι δημοσιογράφοι έχουν πάντα την ελευθερία να είναι επικριτικοί απέναντί μας, αλλά τα θεσμικά όργανα και από πλευρά του ε, δυσκολεύονται πολλέ φορέ να κάνουν την αυτοκριτική τους. Αν την έκαναν λίγο περισσότερο, μπορεί να βελτιωνόντουσαν λίγο ε, τα πράγματα. Όπως σα έλεγα, τα θεσμικά όργανα έχουν ανάγκη να κάνουν ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς το ευρύ κοινό, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και όλες οι πληροφορίες οι οποίες διαβιβάζονται, όπως σας έλεγα, θα πρέπει να στοχεύουν στο χρήστη και όχι σε αυτόν που την αποστέλει, δηλαδή στα θεσμικά όργανα. μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα κατ' εμέ και δεν είναι μόνο θέμα του να κάνει κάποιος κριτική ή να μην είναι επικριτικός. Μπορούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνία και ελπίζω να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στο υψηλότερο επίπεδο για την επικοινωνία μας για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Το... Καταλάβαμε ότι είστε δημοσιογράφος. Οι δημοσιογράφοι πάντοτε μιλάνε για το δημοκρατικό έλλειμμα. Σας παρακαλώ θερμά λοιπόν να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την έκφραση στην έκθεσή σας, διότι είναι ατέριαστη πλέον. Έχετε εδώ φτάσει, έχετε, ε, δουλεύετε σε ένα σώμα εδώ όπου δεν υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα. Πιστεύω ότι συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα, εργαζόμαστε υπεύθυνα και κάνουμε περισσότερο έργο από ό,τι ορισμένα εθνικά κοινοβούλια. Εάν ήξεραν ορισμένοι Γερμανοί συνάδελφοί μου, εθνικοί βουλευτές δηλαδή, τι τραβάμε εμείς εδώ, πόση δουλειά κάνουμε και πόσες ώρες μουχθούμε, πιστεύω θα τραβούσαν τα μαλλιά τους. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, αυτές τις απέσιες, ε, την απέσια αυτή ορολογία δημοκρατικό έλλειμμα, μην τη χρησιμοποιήσετε. Λέτε ότι δεν έχουμε επίτροπο επικοινωνίας. Εγώ σε αυτό θα απαντούσα το εξή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν υπάρχει τέτοιος επίτροπος, ο οποίος θα εισχολεί το μόνο με την επικοινωνία. Ξέρω ότι τον τομέα αυτόν τον έχει η κυρία Ρέντιν και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι έχει επικοινωνία και πολίτες με ποιον θα επικοινωνεί ο, επικοινωνών, ο Επίτροπος της Επικοινωνίας. Με τους πολίτες βεβαίως, με την κοινωνία των πολιτών. Άρα λοιπόν πολύ σωστά συνδυάζονται αυτές οι δύο αρμοδιότητες. Είμαι λοιπόν πραγματικά ευγνώμων που έχουμε μια εξαιρετική Επίτροπο η οποία επιτελεί ένα θαυμάσιο έργο και ό,τι έχει κάνει νομίζω ήταν ιδιαίτερα επιτυχές δεδομένου ότι συνδέει το έργο της επικοινωνία και πολίτες. Επίσης, ε, όσον αφορά τώρα η, τη δημόσια τηλεόραση, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, Πρόσφα... Ε, σύντομα θα έχουμε μια έκθεση του κυρίου Μπέλε, του συναδέλφου μας, με το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ καλά το δικό σας θέμα. Αλληλοσυμπληρώνονται οι δύο εκθέσεις. Τώρα, πολλοί συνάδελφοι ήταν στο παρελθόν επιφυλακτικοί ε, για όλη την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς τώρα έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε το streaming που μπορεί κανείς να παρακολουθεί στις συνεδριάσεις. Ε, πολλοί χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και πολλοί όχι. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ προχωρημένοι και πολύ προοδευτικοί. Έχουμε εξυγχρονιστεί ιδιαίτερα. Ε, μήπως λοιπόν καλό θα ήταν να οργανώσουμε ένα σεμινάριο για τους συναδέλφους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλες αυτές τις τεχνολογίες. Ε, πιστεύω ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο. Το θέμα είναι πώς θα περάσει το μήνυμά μας, όχι για τα θεσμικά όργανα, αλλά για το τι κάνουμε εμείς εδώ, στην ψυχή της Ευρώπης. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εντωμεταξύ έχει γίνει θύμα της δικιάς της επιτυχίας. Θα πρέπει λοιπόν ίσως να διοργανώσουμε μία ακρόαση με τίτλο «Τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση». Ε, ε σήμερα Εάν δείτε τα παιδιά σας, την επόμενη γενιά, τα θεωρούν αυτονόητο ότι υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι ποτέ δεν έχουν δείξει το διαβατήριό του όταν περνάνε τα σύνορα. Για αυτού είναι αυτονόητο ότι δεν έχουμε ελέγχου ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο. Λοιπόν, έχουμε ε, ε, σημειώσει τέτοιες επιτυχίες και αυτούς τους θησαυρού πρέπει να τους διαφυλάξουμε. Καλό λοιπόν πιστεύω ε, θα ήταν να προβάλλουμε καλύτερα τις επιτυχίες μας βοηθώντας και την κυρία Ρέντινγκ. Προχωρούμε στον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πιστεύω ότι είναι μια φιλόδοξη έκθεση, ένα φιλόδοξο έργο αυτό που έχετε αναλάβει και πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να το ολοκληρώσουμε πολύ ε, ικανοποιητικά. Αυτό που θα θέλαμε βεβαίως είναι να έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αυτό θα ήταν ε, ο επιθυμητός στόχος. Πολλά ε, προγράμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, αυτή την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, όπως το DrySat, όπως οι, ευρωπαϊκά, οι ευρωπαϊκές εκπομπές, να τα προωθήσουμε περισσότερο, και οι πολιτικοί μας πάντοτε εκτιμούν ιδιαίτερα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορεί να είναι πολύ ωραία και καλά αυτά τα προγράμματα. Αν όμως δείτε πώς είναι οι αποδέκτες, είναι αρκετά λίγοι. Δυστυχώς ε, δεν έχουν την ε, ακροαματικότητα την οποία θα θέλαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υποβάλουμε πολύ συγκεκριμένα ε, προγράμματα πετραδάκι πετραδάκι θα μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής ε, δημόσιας γνώμης. Συμφωνώ και εγώ με την ε, Πρόεδρο ότι καλό είναι που δεν έχουμε επίτροπο επικοινωνίας, διότι η επικοινωνία είναι έργο του καθενός μας. Και ε, κάθε ένας είναι υπεύθυνος να επικοινωνήσει μέσω του έργου του δεν πρόκειται μόνο για μια μικρή ταινία, ε, βίντεο ή μια ταινία μικρού μήκους ή ένα προγραμματάκι σε βίντεο. Δεν πρόκειται μόνο περί αυτού. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε, να φτάσει το μήνυμά μας, το ουσιαστικό, στους πολίτες μας και να μην ε, χάνονται οι δραστηριότητες μας ε, στα περιφερειακά και εθνικά κοινοβούλια, να μην πνίγονται δηλαδή. Τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ε, στη Γερμανία έχουν μια συγκεκριμένη δομή βάσει της οποίας λειτουργούν και στην, στο Ενωμένο Βασίλειο. Και λειτουργούν βάσει του ενός νομικού πλαισίου δημοσίου δικαίου. Δεν θα πρέπει όμως να παραγνωρίζουν και την ευρωπαϊκή πτυχή στο νομικό τους πλαίσιο. Η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να θεμελιωθεί και να παγιωθεί σταθερά όταν επιβάλλουμε την ευρωπαϊκή πτυχή σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή σε όλα, σε όλα τα προγράμματα ή σε όλα τα θέματα τα οποία προβάλλονται από, τη μέσα, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην παραβλέπετε και παραλείπετε η ευρωπαϊκή διάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση σε όλους τους τομείς των μέσων ενημέρωσης και δι στην εκπαίδευση των δημοσιογράφων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι δημοσιογράφοι αυτοί να έχουν το πλεονέκτημα της επιμόρφωσης σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκά θέματα, διότι ενισχύεται και η, η, συνεργασία η, μεταξύ ευρωπαϊκής και εθνικής ε, πολιτικής ή ευρωπαίων και εθνικών δημοσιογράφων. Θα, θα πρέπει βεβαίως ε, σε εθνικό επίπεδο να προβάλλονται οι τα, τα, τα, θέματα τα οποία αφορούν την εθνική κοινωνία, τους πολίτες, αλλά πολλές φορές λείπει τελείω η, ευρωπαϊκή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως λέγαμε πριν, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έχουμε το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, το οποίο μας κάνει όλους πάρα πολύ υπερήφανος, διότι είναι θαυμάσιο και πιστεύω ότι δείχνει πολύ σωστά την ε, κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να έχει το νομικό πλαίσιο δημοσίου δικαίου για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, δημόσιας ενημέρωσης, τα δημόσια μέσα. Πολλές ε, φορές ζητούμε το, τα δημόσια μέσα ενημέρωσης να μας προβάλλουν πολύ περισσότερο και μας λένε από τη δική τους πλευρά ότι δεν μπορούμε διότι υπάρχουν νομικοί περιορισμοί. Πρέπει λοιπόν αυτά να ξεπεραστούν. Η κυρία Τρούπελ. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη και την ευρωπαϊκή συνείδηση, έχω ένα σχόλιο. Ε, ήμασταν στη οι πέρσι, ένα μέρος της ε, Επιτροπή Πολιτισμού, και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στη Στοχόλμη μας είπε ότι το 2010 στη Σουηδία θα έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Μα τι είναι αυτό. Κοιταχτήκαμε όλοι μεταξύ μας και μας λέει ακριβώς αυτή την αντίδραση ήθελα να δω σε εσά. Βεβαίως δεν είναι ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά εμείς θεωρούμε και τις ε, εθνικές εκλογές ως ευρωπαϊκές, διότι έτσι μπορούν οι πολίτες μας να εκφράσουν τη γνώμη τους και επί ευρωπαϊκών θεμάτων, ανάλογα με τα κόμματά τους δηλαδή. Αυτό όμως δεν είναι προφανές σε όλες τις χώρες και αυτό είναι μια πτυχή του ευρωπαϊκού προβλήματος. Μπορούμε να γράψουμε ατελείωτες εκθέσεις για το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. κλπ. Αλλά ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση. Εμείς δεν είμαστε τα Ηνωμένα Έθνη της Ευρώπης, εμείς είμαστε αυτή, το ειδικό μείγμα εθνικής και υπερεθνικής δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική έλλειψη γνώσεων και ουσιαστικής ενημέρωσης ε, των δημοσιογράφων για την ουσία της ύπαρξής μας. Αυτό το διαπιστώνουμε συνέχεια, πολλές φορές. Όταν ρωτάνε περί τίνος πρόκειται, τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί δημοσιογράφοι συνεχώς ρωτάνε και με τίτλους μεγάλους, π.χ. τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους. Και λένε συνέχεια ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα και δημοκρατικό έλλειμμα, μια καραμέλα δηλαδή την οποία επιπηλίζουν συνέχεια. Πολλοί ε, και πολιτικοί το ισχυρίζονται αυτό και λένε ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο μπορούμε να το υπερνικήσουμε, να το ξεπεράσουμε εάν διαλύσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, δηλαδή πλήρης ε, σύγχυση. Εμείς δεν έχουμε πολιτική πλειοψηφία για να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις ε, τέτοιες περί ε, ομόσπονδης Ευρώπης, περί Ηνωμένων Πολιτειών ε, της Ευρώπης. Δεν έχουμε ούτε την αρμοδιότητα ούτε και τη διάθεση να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά υπάρχει αυτή η ενημέρωση, αυτή η παρουσίαση του μιας τέτοιας πλευράς από τον τύπο. Είναι ένα είδος δηλαδή δημοσιογραφικού κουτσομπολιού, όπως λέμε στη Γερμανία, το οποίο πιπιλίζεται συνέχεια και ε, αναφέρεται συνέχεια και δει στις πρώτες σελίδες και στα κύρια άθρα. Δημοκρατικό έλλειμμα σε εισαγωγικά συνέχεια εμφανίζεται. Άρα λοιπόν, θα πρέπει η το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο να συγκεραστούν, να συγκλίνουν και θα πρέπει οι δημοσιογράφοι, και τα δημοσιογραφικά μέσα να εξηγήσουν πώς τα δύο αυτά τα επίπεδα συνεργάζονται, συγκλίνουν, συνενούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε ποια είναι η πολιτική θέση του καθενός και σε τι στηρίζεται. Ε, δεν είναι δυνατόν λοιπόν ε, να μιλάμε για Ηνωμένε Πολιτείε ε, τη Ευρώπη, σαν τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής, εκτός από μερικέ ε, πολιτικές ομάδες, ας πούμε, όπως το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα που αναφέρεται σε αυτό. Αλλά αυτά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Δεύτερο θέμα, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, για τους δημοσιογράφους και τα νέα τεχνολογικά μέσα, όπως το ίντερνετ, Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο στη Γερμανία ε, που αφορούσε τις επιθυμίες και τις προσδοκίες των πολιτών και έλεγε το άρθρο ότι πρώτη φορά έγινε μία διαβούλευση ε, στο διαδίκτυο για τις επιθυμίες, να καταγραφούν οι επιθυμίες των Ευρωπαίων πολιτών. Και όμως αυτές οι βλακίες αναφέρονται συνέχεια στον τύπο, ενώ γίνονται συνέχεια ε, online consultations, δηλαδή ε, διαβουλεύσεις και συζητήσεις στο διαδίκτυο για το ένα και το άλλο θέμα. Δεν είναι λοιπόν ε, παραδεκτό ότι την πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2009 έγινε μία διαβούλευση στο διαδίκτυο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπάρχουν άπειρες συζητήσεις που γίνονται μέσω του ίντερνετ νέοι, ομάδες νέων στα πανεπιστήμια και μέσω του ραδιοφώνου και μέσω του διαδικτύου υπάρχουν ε, ειδικέ ομάδες ενδιαφέροντος οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Υπάρχουν θαυμάσιες ιδέες λοιπόν με, με την τεχνολογία αυτή για το τι μπορεί κανείς να κάνει για να μεγαλώσει την πρόσβαση και την ακροαματικότητά του και την διάδοση του μηνύματος. Τα είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάμιμπολ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν σχεδόν με όλα. Όσον αφορά τη γενικότερη πολιτική μας θέση, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει ε, αδιαφορία μόνο για τις ευρωπαϊκές εκλογές, αλλά και αλλού, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να δει κανείς γενικότερα στο δυτικό κόσμο μια τέτοια στάση. Μια γενικότερη απογοήτευση, απογοήτευση αν θέλετε, με το, με το πολιτικό σύστημα, με τον τρόπο που λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα. Και αυτό φαίνεται, αποκρισταλώνεται στην αδιαφορία των ε, πολιτών. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Συμφωνώ με την κυρία Πάκ ότι πρέπει να σταματήσουμε πλέον να μιλάμε για το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα. Πάντως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα όσον αφορά την συμμετοχή των πολιτών. Ζήτημα το οποίο δεν εντοπίζεται μόνο στην Ευρώπη. μένω σας μην επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στο ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι γενικότερο και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε έναν τρόπο για να το αντιμετωπίσουμε. Υπό το φως όμως του γεγονότος αυτού, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ευρώπη προκειμένου να βελτιώσουμε τη δική μας την κατάσταση. Ω δημοσιογράφο, εσεί θα το γνωρίζετε πολύ περισσότερο και διστάζω να το πω αυτό σαν δημοσιογράφο. Πάντω, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερε ιστορίε, αν θέλετε, πολύ περισσότερο από ό,τι κάνουμε. Ένα από του λόγου ε, που δεν αναφέρεται συχνά σε άρθρα η Ευρώπη είναι ότι δεν παρουσιάζουμε τελικά τον εαυτό μα με ενδιαφέροντα τρόπο. Και σαφώ αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν πρέπει κανεί να αντιμετωπίσει 27 κράτη-μέλη, τρία θεσμικά όργανα και όταν πρέπει να εργαστεί κανεί με μια διάρθρωση σαν αυτή την οποία έχουμε εμεί. Είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανεί ανθρώπινο πρόσωπο σε όλο αυτό το οικοδόμα και να το καταστήσει ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δυστυχώ αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι παρουσιάζουμε τα πράγματα πολύ διοικητικά, πολύ θεσμικά και οι πολίτε δεν μπορούν να ταυτιστούν με κάτι τέτοιο. Και επίση υπάρχει και ένα πρόβλημα εθνικών μέσων ενημέρωση. Και το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδεχομένω το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει τη χειρότερη κατάσταση, αλλά δεν είναι η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η μόνη χώρα που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, αρνητική στάση δηλαδή των εθνικών μέσων ενημέρωση. Νομίζω ότι σαφώ μπορούμε να μιλάμε για το BBC και για άλλα δίκτυα, αλλά όλα αυτά αποτελούν τμήμα μόνο του προβλήματο. Και να πω επίση ότι για το ζήτημα αυτό. Το BBC έχει ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Record Europe, μια, ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα που συζητούν τα ευρωπαϊκά θέματα. Και δύο εκατομμύρια είναι οι τηλεθεατές του προγράμματος αυτού στην Ομένο Βασίλειο, το οποίο θα μου πείτε ότι δεν είναι ένας τεράστιος αριθμός. Παρ' όλα αυτά είναι ένας αξιοπρεπής, αν θέλετε, αριθμός. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κάποιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν αυτά τα δύο εκατομμύρια ανθρώπων, ακόμα και στην Ευρωσκεπτική, Ευρώπη, ε, Βρετανία, με συγχωρείτε, που παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ακριβώ το ενδιαφέρον αυτό που υπάρχει. Και αυτό μπορεί να γίνει κυρίω σε εθνικό επίπεδο, γιατί όπω ε, είπε η κυρία Τρούπελ πάρα πολύ σωστά, πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια μεμονωμένων κρατών μελών. Δεν είμαστε ακόμα ένα υπερεθνικό κράτος. Τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά από ένα κράτο στο άλλο. Για παράδειγμα, ε, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ, μάλλον δεν μου αρέσει καθόλου ότι μιλάμε για πολίτες, citizens. Κανείς στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναφέρεται στους πολίτες κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένω, κάθε φορά που ακούω τον όρο European citizens, ε, Ευρωπαίοι πολίτες, αυτό μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν αναφέρει κανεί τον όρο European Citizens, κατευθείαν οι άνθρωποι να τριχιάζουν και ουσιαστικά χάνουν κάθε ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσελκύσουμε ουσιαστικά το ενδιαφέρον. Και κάτι ακόμα. Όσο μονομένοι ευρωβουλευτέ, έχουμε κι εμεί μια ευθύνη. Ιδίω στην πρόσβαση που έχουμε εμεί στα νέα μέσα. Πάντα λέμε ότι κάποιο άλλο θα πρέπει να κάνει τη δουλειά μα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Έχουμε πρόεδρο πλέον, έχουμε και είπα το αρμοστή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι εμεί μπορούμε να κάνουμε οι ίδιοι πολύ περισσότερα πράγματα. Εμεί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα νέα μέσα ενημέρωση, ενδεχομένως να δυσκολευόμαστε να έχουμε πρόσβαση τεχνικά τεχνικά μέσα ενημέρωσης, παρόλα αυτά σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή πρόσβαση και να πρόκειται σε εμά τελικά να κάνουμε διάφορα πράγματα, να λάβουμε ευθύνε και πρωτοβουλίες οι ίδιοι για να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Μπαντία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αν ήταν ε, σημαντική και περίπλοκη η προηγούμενη έκθεση, αυτή πια ξεπερνάει τα εξκαμένα. Ε, ένα-δυο πράγματα, γιατί ήδη ακούστηκαν πολλά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λόκεγκάρντ για τα σχόλιά του και ο ίδιος επέμεινε στο ότι θα πρέπει να επικοινωνούμε περισσότερο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα και πρέπει να ξέρουμε και τι πληροφορίε διαβιβάζουμε πολλές φορές ακούγεται ότι κάνουμε προπαγάνδα με την επικοινωνία και επομένως οι πολίτες ούτε καν ενδιαφέρονται και ούτε τους δίνεται εντύπωση ότι προσπαθούμε να τους επικοινωνήσουμε. Τους δίνεται εντύπωση ότι προσπαθούμε να τους πουλήσουμε κάτι. Ε, λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει επιτυχία στα σκάνδαλα. Οτιδήποτε είναι ε, τέτοιας μορφής που λέτε ε, έχουμε όλοι μια κουλτούρα του όχι. Οτιδήποτε πάει αντίθετα σε κάτι πουλάει πολύ. Και επομένως το να κάνουμε κάτι υπέρ κάποιου πράγματος στοιχίζει πολύ περισσότερο. Επίσης μας είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, εθνικών βουλευτών, των περιφερειακών βουλευτών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εγώ συμφωνώ απολύτως και μάλιστα στη χώρα μου προσπαθώ να τα οργανώσω λίγο καλύτερα τα πράγματα και πάντα χρησιμοποιώ ως παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ ξέρω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όταν ξεκινάει η συζήτηση μιας οδηγίας εδώ, ξεκινάει ταυτόχρονα συζήτηση σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι εκπληκτικό. Από εκεί και πέρα, το κατά πόσον οι πολίτες θα βλέπουν με καλύτερο μάτι την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου σας απαντά απευθεία. Το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο και ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Νομίζω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενδιαφέρονται για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτοί πηγαίνουν στο Συμβούλιο. Όταν υπάρχουν Συμβούλιο, όταν υπάρχουν συνεδριάσει του Συμβουλίου, όλο ο τύπο είναι εκεί. Εδώ έχουμε αυτούς, εκεί συγγνώμη, έχουμε αυτούς που θεωρεί ο τύπος ότι έχουν την εξουσία, αυτούς που δίνουν τις διαταγές και τις εντολές και το να έρθουν εδώ ε, τους στοιχίζει πολύ και τους στοιχίζει και πολύ γιατί δεν γνωρίζουν τα θέματα που συζητάμε εδώ. Ε, δεν γνωρίζουν τα θέματα γιατί συνήθως συζητάμε πιο τεχνικά ζητήματα και νομίζω ότι στη χώρα μου λίγο πολύ αυτό συμβαίνει. Ο τύπος αγνοεί κάποια πράγματα, αγνοεί την ουσία των θεμάτων που συζητάμε και επομένως τους δυσκολεύει και δεν τους ενδιαφέρει γιατί ακριβώς δεν το γνωρίζουν. Όταν ε, εξετάζαμε τα θέματα αυτά και κάναμε τις ακροάσεις των επιτρόπων ε, πριν από κάποιες εβδομάδες, ήρθε ένα ε, κάποιοι, ήρθαν κάποιοι εκπρόσωποι ενός ε, καθημερινού προγράμματος ε, στην ε, Ισπανία. Ε, ο δημοσιογράφος που ήρθε ήξερε όλα τα θέματα που συζητούνταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πρόγραμμα το οποίο έγινε βάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκε η τηλεθέαση του προγράμματος το οποίο ήδη τη μεγάλη μεγάλης θεαματικότητα στην Ισπανία. Συμφωνώ επίσης με τα όσα ακούσαμε εδώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ξεχάσουμε πλέον αυτό το θέμα του δημοκρατικού ελλείμματος. Γιατί πιστεύω ότι δεν είναι αλήθεια. Εμείς εκλεγόμαστε άμεσα από τους πολίτες. Το Συμβούλιο, ε, δεν μπορεί να μιλάμε και για το Συμβούλιο για Δημοκρατικό Έλλειμμα, διότι και αυτοί ε, είναι εκλεγμένοι απευθεία από τους πολίτες. Πρέπει να εξηγούμε λίγο τα πράγματα όπως είναι και να μην τα μπλέκουμε μόνοι μας. Και επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε περάσει τόσα χρόνια ε, για τη συζήτηση επιθεσμικών θεμάτων. Είτε αυτό ήταν το Σύνταγμα, είτε το οτιδήποτε. Τόσα χρόνια επιβαρύνουμε τους πολίτες με όλα τα θεσμικά μας ζητήματα. Και όντως, αυτά δεν τους ενδιαφέρουν. Κανένας δεν αντέχει 50 χρόνια συζήτηση για το σύνταγμά του ή και για την περίπτωσή μου για την Καταλωνία, για το μικρό μας ε, σύστημα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα έχουμε λίγο κατανό θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα και στο κεφάλι μας και να δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό και πού μπορούμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία και να παρουσιάσουμε και ε, συγκεκριμένες ιδέες που θα μας βοηθήσουν να πάμε λίγο παραπέρα. Ευχαριστώ. Μου είπε ο μου ότι είναι, ο οποίος είναι και Βρετανός υπήκος και μου λέει δεν, δεν είμαι Βρετανός υπήκος, είμαι υπήκονος της ε, αυτού μεγαλειότητος. Του βασιλείου δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, ε, κάθε χώρα έχει τις παραδόσεις της, ε, έχει τα πιστεύω της, ε, δεν μπορούμε όλοι να αισθανόμαστε το ίδιο, αλλά πιστεύω ότι και ο γραμματέας μας αισθάνεται Βρετανός ε, ε, υπήκος του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και Ευρωπαίος. Αλλά ας μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να πω στον εισηγητή ότι θα λάβει το λόγο μετά την Κομισιόν. Θέλει η Κομισιόν να παρέμβει. Σας ευχαριστώ, Adam Watson από την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μέσους Ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησα τη συζήτηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει την κατεύθυνση που παίρνει η συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Mr. Lockegaard, please. Okay. Sure. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Lockegaard. Ευχαριστώ για όλες τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και όλα τα σχόλια που έγιναν. Αυτή η ζωντανή συζήτηση έδειξε πόσο καυτό είναι αυτό το θέμα και ενδιαφέρον. Θα συνοψίσω τις παρατηρήσεις. Δεν θα να απαντήσω λεπτομερώς. Λοιπόν, το δημοκρατικό έλλειμμα. Ίσως με παρανοήσατε λίγο για το τι εννοούσα δεν λέω ότι εδώ υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα, διότι εδώ έχουμε ένα πλεόνασμα <laughs> δημοκρατίας, όχι έλλειμμα. Θέλω απλώς να το αναφέρω αυτό ως ε, τον όρο αυτό σημείο εκκίνησης για να πω ότι ε, όλοι οι πολιτικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην ε, περαιτέρω ανέλυξη ε, της δημοκρατίας. Ε, εμείς ως δημοσιογράφοι ε, πρέπει να θέτουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Άρα λοιπόν καθήκον μας είναι να περνούν οι απόψεις ε, των πολιτών στα ε, αρμόδια και ενδιαφερόμενα, στους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς, στους πολιτικούς, στους ηθήνοντες. Εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε ένα σωρό μέσα στη διάθεσή μας. Έχουμε ε, πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δουλεύει ε, βέλτιστα αυτή η μηχανή. Δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η, η επικοινωνία, είναι και παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο αφορά την επικοινωνία μεταξύ των πολιτικών φορέων. Ο καθένας ε, βέβαια από εμά προέρχεται από μια πολιτική κουλτούρα και αυτό είναι διεθνές φαινόμενο. Μας ε, πάρουμε παράδειγμα αυτό που είπε ο Βρετανός ε, πίκος, ο φίλος μας μόλις τώρα. Ακριβώς όλοι έχουμε ένα παρελθόν, μια κουλτούρα την οποία έχουμε ενστερνιστεί. Και γι' αυτό εμείς ε, οι δημοσιογράφοι που εκπροσωπούμε την κοινή γνώμη πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους ορισμούς. Δηλαδή πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τις δύο πλευρές, ε, ε, την πηγή με τους αποδέκτες. Αυτό πρέπει να είναι το καθημερινό μας έργο. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά το Μάρτιο της συνεδρίασή μας θα έχουμε το σχέδιο της εκθέσεως για να δούμε τι έχει συμπεριλάβει ο εισηγητής από τις ιδέες μας και τα σχόλια μας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, λίγη συνεδρίαση, έχουμε λάβει και τα πρακτικά. Αν δεν έχετε καμία αντίρρηση, θα θεωρήσω τα πρακτικά ως εγκρισέντα. Πιστεύω ότι θα τα έχετε όλοι διαβάσει.